Αγαπητοί συνάδελφοι, στα γαλλικά, στα ισπανικά και στα ιταλικά και στα αγγλικά. Καθίστε παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Και να είστε και ήσυχοι. Για να ξεκινήσουμε το συντομότερο. Πρέπει να στήσουμε συγνώμη για την ε, πλέον ασυνήθιστη αυτή κατάσταση από τον οριστέντα επίτροπο. Ήταν εντελώς απρόβλεπτο, έκτακτο. Τόσα χρόνια στο κοινοβούλιο πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Στην Τενερίφη είχαμε μπλάκα ούτε 9 ώρες. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έζησαν στο πλήρε σκοτάδι την Κυριακή την προηγούμενη. Φοβήθηκα λοιπόν. Λέω κατάρα είναι αυτή. Ευτυχώς όμως ε, εδώ χρειάστηκε πολύ λιγότερος χρόνος από ό,τι φοβόμαστε για να λυθεί το πρόβλημα. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά τους κλητήρες μας, οι οποίοι έκαναν πάντο δυνατό για να είναι έτοιμοι σε λιγότερο από μισή ώρα αυτή η αίθουσα. Τους ευχαριστούμε θερμά. so And now if you, if you... Και τώρα, αν συμφωνείτε, Πίτρο ε, στο μέσο της απάντησης ε, προς την κυρία Μπρίκμο νομίζω ότι θα ήταν καλό να δώσω το λόγο στην κυρία Πρισκμό για να κάνει τη δεύτερη, την Μπρικμό να κάνει τη δεύτερη της ερώτηση, γιατί ολοκλήρωνε την απάντησή του ο Επίτροπος. Ναι, ευχαριστώ και εγώ τις υπηρεσίες, λέει κυρία Μπρικμό. Ελπίζω να μην ε, ήταν ένα είδος λογοκρισίας, γιατί άκουσα και εκτιμώ την απάντησή σας αγαπητέ ε, Πίτερο Θέλω όμως ε, να επιστρέψω την προσοχή σας σε δύο παραδείγματα. Την ε, σύλληψη μιας οικογένειας Οιγούρων, που είναι μια μειότητα που δέκεται στην Κίνα. Η σύλληψη έγινε στην Βελγική Πρεσβεία στο Πεκίνο και Τρει μήνε μετά δεν ε, έχουν αντιδράσει για την επανένωση οικογένεια στο Βέλγιο. Οι βελγικέ αρχέ επίση, ε, συνεργασία του Βελγίου με το Σουδανικό καθεστώ για την ε, σύλληψη και έκδοση Σουδανών υπηκών που είναι πολύ πιθανό ότι θα υποστούν βασανιστήρια και θα διωθούν αυτοί. Λοιπόν, είναι η αντίληψη που έχετε για την εξαγωγή των πρότυπων και ευρωπαϊκών αξιών ε, και σκεφτόμουν ειδικώ ε, τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης Προστασία των ε, Δικαιωμάτων Ισότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη. Ελπίζω το άρθρο 2 για την προστασία λοιπόν των ελευθερών και των δικαιωμάτων να ε, το λάβετε υπόψη ε, και να το τηρήσετε ως Επίτροπος ε, στις δεσμεύσεις σας και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Μπρικμό. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι είμαι αποφασισμένος να γίνει σεβαστό το άρθρο 2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε να εξαγάγουμε τα πρότυπά μας. Δεν υπήρξε όμως για να σας διορθώσω σύλληψη στη Βελγική Πρεσβεία του Πεκίνου. Απλά ε, επειδή ήταν ε, σε εξέλιξη διαδικασία επανένωσης, ε, απλά μεταφέρθηκε αυτή η οικογένεια και μάλιστα θα πάρουν διαβατήριο από τις κινέζικες αρχές. Εμείς θέλουμε να υπάρξει επανένωση οικογένειας, είμαστε σε συνεχή επαφή με τις κινέζικες αρχές και με την οικογένεια, τόσο εδώ όσο και στην Κίνα, στο Σινγκιάν και ξέρετε ότι συχνά παρεμβαίνουμε, διότι η πολιτική του Βελγίου σε θέματα διεθνή είναι γνωστή ε, και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι παντού προωθούμε τις αξίες αυτές και στο πλαίσιο του ΕΕ και αλλού και μιλώ και για τη μεταναστευτική πολιτική και για άλλες πολιτικές όπου θέλουμε να γίνονται πλήρω σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αξίες μας και αυτό να φαίνεται σε όλες μας τις πολιτικές. Τώρα έχουμε τον εκπρόσωπο της ομάδας ID, ε, κύριο Τόμ Φαντεντρίσε. Καλημέρα σας ε, κύριε Ρέντερς. Ε, θα πρέπει να ελέγξετε την λειτουργία του κράτους ε, δικαίου. Βλέπουμε όμως πως στο Βέλγιο το μισό του συνταγματικού δικαστηρίου είναι πολιτική και κατέληξε ενώπιον του δικαστηρίου αυτού το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας ενώπιον ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Και τι βλέπουμε εκεί πέρα, μπορούν να εξαγοραστούν ε, οι ποινές οι οποίες επευλήθησαν για φορολογικές απάτες. Τα ΟΟΗΕ επίσης ασκεί κριτική για τις συναλλαγές με την ε, Λιβύη και την σχετική διαφθορά. Και ξαφνικά σταματάει η έρευνα αυτή ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να γίνει η ακρόασή σας, οποία σύμπτωσης. Έχουμε βεβαίως και την σχετική έκθεση της κρατικής ασφάλειας. Μα μετά από όλα αυτά πώς να σας εμπιστευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την προστασία του δημοκρατικού κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, η απάντησή σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, ερώτησή σας. Θα ήθελα να πω το εξή. Είπα στην εισαγωγή μου τα όσα, αφορά, τα, τα όσα αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα ήθελα να πω ότι θα δώσω πραγματικό αγώνα για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου εντός της ε, Ένωσης και εκτός της Ένωσης. Και είναι σημαντικό να πω πως ε, θα προχωρήσω στην κατάρτιση μιας ετήσιας έκθεσης για το κράτος ε, δικαίου, ένα νέο μηχανισμό, χωρίς καμία διακριτική μεταχείριση του χ του Δηλαδή και όσον αφορά το Βέλγιο θα γίνουν μια σειρά παρατηρήσεις και νομίζω ότι η καλύτερη απόδειξη για την βούλησή μας για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου ε, είναι αυτή. Εδώ και τρία χρόνια πρότεινα να γίνει μια τέτοια έκθεση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ε, ενώπιον του Συμβουλίου, με και είπα ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται για κάθε ε, κράτος μέλος, όχι μόνο εκεί όπου είναι εμφανή τα προβλήματα. Τώρα, για τους δικαστές ε, στο Βέλγιο, ο ορισμός τους είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία, όπως ε, ξέρετε. Υπάρχει ένα ειδικό συμβούλιο για την δικαιοσύνη Αυτά τα πράγματα γίνονται και σε πολλέ ε, άλλε χώρε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ε, ένομη τάξη του Βελγίου και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι έδωσα συγκεκριμένη απάντηση για το θέμα αυτό στην εισαγωγή μου. Σας ευχαριστώ. Έχετε ξανά το λόγο για ένα λεπτό. λέτε ότι θα υπερασυστείτε τα αστικά δικαιώματα, ένα ε, εκ των οποίων είναι η ελεύθερη γνώμη. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να είναι απαραβίαστο, ανήκει στον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε ασυνήθιστες και ε, ανεξέλεγκτες μαζικές μεταναστευτικές ροές. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν είναι ότι παραβιάζεται η ελευθερία γνώμης όποιου καταδικάζει αυτήν την πολιτική. Ταυτόχρονα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίε για να ποινικοποιηθεί η ελεύθερη γνώμη επί του θέματος αυτούς. Ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως το Facebook στρατολογούνται για να λογοκρίνουν. Αυτό δεν έχει δε μία σχέση με ρατσισμό, hate speech κτλ. αλλά με περιορισμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας γνώμης. Ποια πρωτοβουλία θα αναλάβετε για να προστατεύσετε την ελευθερία λόγου και να την ερμηνεύσετε όσο δυνατόν πιο διασταλτικά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρεντέρς, Βεβαίω ε, είμαστε υπέρ τη ελευθερία του τύπου και του κάθε πολίτη να εκφράσει την άποψή του και για την ε, μετανάστευση βεβαίω. Ε, Πολλέ και διαφορετικέ νόμου. Όχι μόνο και στο Εθνικό μα Κοινοβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύονται ε, διαφορετικέ απόψει. Αλλά μετά από εκεί υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορούμε να περάσουμε στον ρατσισμό όπω το είπατε κι εσεί. Υπάρχει μια πραγματική διαφορά μεταξύ ε, των διαφόρων κανόνων ή του ανοίγματο ή μη στη μετανάστευση και της επίθεσης ε, στον μετανάστη ή στους αλλοδαπούς με βάση τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Θα κάνουν τα πάντα λοιπόν για να υπάρχει ένα σωστό όριο μεταξύ ε, της ελεύθερης άποψης που πρέπει να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα αλλά πραγματικός ρατσισμός ή πραγματικά ε, ποινικά δικήματα ε, που αφορούν τον ε, ρατσισμό είναι κάτι άλλο. Και πάλι αυτό είναι δουλειά όμως των δικαστών για να το αποφασίσουν. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον εκπρόσωπο του ECR. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να συλλάβουμε εγκληματίες εντός της Ένωσης. Συγκεκριμένα με αυτό το ένταλμα μπορούν τα εθνικά συστήματα να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα και να λειτουργήσουν καλύτερα. Το προηγούμενο κοινοβούλιο και η θητεία έχουν εργαστεί επί ετών σε μια μεταρρύθμιση του συστήματος αυτού αλλά ε, για να μην χρησιμοποιηθεί με τρόπο δυσανάλογο. Έτσι θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να λειτουργήσουν, να ζητήσουν την σύλληψη σε ένα άλλο κράτος μέλος ε, με τρόπο ειλικρινή και αναλογικό. Κύριε Ρέντερς, μπορείτε να διαβεβαιώσετε το κοινοβούλιο μας πως η Κομισιόν θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Τέλμα Σύλληψης να λειτουργήσει σωστά και όλα τα μελλοντικά μέτρα για δικαστική συνεργασία θα παραμείνουν στον αντικειμενικό του σκοπό και δεν θα είναι αντικείμενο κατάχρησης, γιατί βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη στο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να καταλύσει ένα άδειο κέλυφος. Σας ευχαριστώ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, ερώτησή σας ε, για το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνεργασία μας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Πρόκειται για ένα success story. Ε, η δυνατότητα δηλαδή που υπάρχει δίωξη των εγκληματιών σε άλλη χώρα. Είναι χρήσιμο λοιπόν, όπως είπαμε, να παραμείνουμε στο μέτρο της αναλογικότητας και να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας των ε, νομικών μηχανισμών και της υπεράσπισης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι πάντα χρήσιμο να επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν, υπάρχει βεβαίως ε, το δικαίωμα της ε, υπεράσπισης αλλά και πρέπει να υπάρχει και μια αποτελεσματικότητα της ε, διαδικασίας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 40 τέτοια εντάλματα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει άρα μια επανεπεξεργασία της οδηγίας αυτής. Όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη, Αναμένω από τις αρχές του επομένου έτους μια αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την λειτουργία της διαδικασίας αυτής. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πρέπει να πάμε δηλαδή σε μια πλήρη και σωστή εφαρμογή των κανόνων και έχουμε όπως είπα και, θέση, και υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΚ που εκκρεμούν σε σχέση με την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Αλλά με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης νομίζω ότι θα προβούμε σε μια σειρά προσαρμογών με τη σύμφωνη γνώμη οπωσδήποτε του Κοινοβουλίου για να προχωρήσει και η Κομισιόν. Οπότε είμαστε υπέρ αυτής της προσέγγισης της ε, αναλογικότητας και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, αλλά νομίζω πως είναι μια σημαντική επιτυχία. Είχαμε 17.000 ε, τέτοιες ε, υποθέσεις. Ε, σας ευχαριστώ. Έχετε άλλο ένα λεπτό. Ε, είπατε πως είναι πάρα πολύ σημαντική αποτελεσματικότητα και στην επιστολή ανάθεσης ε, καθηκόνων λέγεται πως η καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών πρέπει να προωθηθεί. Γι' αυτό θα ήθελα μια, να σας κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση. Το πώς θα προωθήσετε δηλαδή την αποτελεσματικότητα. Παραδείγματο χάρη ε, όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων ε, που λαμβάνονται όταν εκπνεύσει η νομοθεσία για την ε, συνεργασία μεταξύ διαφόρων θεσμικών οργάνων. Θα ένα παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το, μου το είπαν και επιτόπου στη Europol και αλλού να έρευνουν και να έχουν όλες αυτές τις δυσκολίες για να λάβουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες. Και ο... είναι αντικείμενό σας και η καλή συνεργασία και εδώ πέρα εντάσσεται και η ανταλλαγή πληροφοριών, την οποία θα πρέπει να διευκολύνεται. Οπότε δεν θα πρέπει μόνο να εστιάζετε στους κανόνες, αλλά να φροντίσετε και για την εύκολη εφαρμογή. Κύριε Ρέντερς, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να πάμε προς μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και η Κομισιόν πρώτα απ' όλα θα εξετάσει την σωστή εφαρμογή όλων των ευρωπαϊκών κανόνων και γεγονός είναι ε, έχετε δίκιο και εγώ είχα πάει στην ε, Europol και άκουσα ότι δεν ήταν τόσο απλό να λάβουν ε, πληροφορίες από τα μέλη της Europol Υπάρχει βεβαίως και η εμπειρία με την Interpol στο διεθνές επίπεδο, αλλά δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει, όπως είπατε, να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες και στην ανάγκη θα προσφύγουμε στο 10 αν δεν υπάρξει η σωστή εφαρμογή. Κατόπιν θα πρέπει να δούμε όλες αυτές τις υπηρεσίες, Eurojust, Europol κτλ. Να δούμε ακριβώς το θέμα και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι δυνατόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να συνεργάζονται και να εφαρμόζουν σωστά τους ε, κανόνες. Και επαναλαμβάνω, να γίνεται αυτό για όλη την ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία. Θα καταβάλουμε λοιπόν κάποιες επιπλέον προσπάθειες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Σας ευχαριστώ και πάλι. Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ε, γύρος ερωτήσεων, ήρθε η στιγμή της Γκουε. Η κυρία Ομπρί έχει τον λόγο. Καλημέρα σας κύριε Ρεντέρ. Σήμερα δεν εκφράζομαι εξ ονοματός μου ούτε εκ μέρους της ομάδας μου της Γκουεντζιέλα αλλά εκ μέρους πάνω από 80 οργανώσεων που αύριο θα δημοσιοποιήσουν μια σαφή έτσι προς την Κομισιόν για μια ευρωπαϊκή οδηγία για το δικαίωμα επαγρύπνησης, επιτήρησης. Μιλάμε για χιλιάδες θύματα ουσιαστικά που ζητούν να, να δικαιωθούν από επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. 2.500 εργαζόμενοι στη Ράνια Πλάτσα που εργάζονται για το Καρφούρ και άλλες επιχειρήσεις. Οι Ιταλοί του Τάρες που ε, υπέστησαν την ρήπανση και ε, Λουμπριζόλ στη Γαλλία, μια ακόμη επιχείρηση που ρηπαίνει. Είπατε ότι δεν αρκεί η εθελοντική δέσμευση ε, και η ε, κινήσεις. Ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να υπάρχει πραγματικά ένα, ε, μια υποχρέωση επαγρύπνησης, ε, vigilance. Δεν είπατε τη λέξη αυτή. Τι θα κάνετε λοιπόν για να σταματήσουν τα φαινόμενα τιμωρησίας των πολυεθνικών. Κύριε Εντέρς, έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ομπρί, Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος ε, στο θέμα αυτό. Ε, σίγουρα θα πλαισιώσω τους καταναλωτές ώστε τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά από τις επιχειρήσεις ε, και τους καταναλωτές. Θέλω να προστατεύσω και τους πολίτες. Θα έχουμε λοιπόν μια οδηγία για τις δράση παράστασης ε, και θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, σε μεγαλύτερη εγρήγορση απέναντι σε τέτοιες παραβιάσεις ε, που πλήττουν τους εργαζομένους επιχειρήσεων τις οποίες αναφέρατε και όπου παρατηρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος, το πρώτο που θα κάνω, αν πρέπει να διαβάσω πάρα πολύ προσεκτικά την πρόταση που θα καταθέσουν αυτές οι οργανώσεις, αν σας κατάλαβα καλά αύριο για την πρόταση οδηγίας αυτή. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα κατά πάσα πιθανότητα να τη συζητήσουμε την πρόταση οδηγίας αυτή εδώ ε, στο σώμα. Καταλαβαίνω ποια αίσθηση ε, υπάρχει, ότι θέλετε να πάμε στο δυνατόν πιο μακριά Δηλαδή ε, να περάσουμε από οικειοθελείς κινήσεις σε υποχρέωση ε, που θα την νομοθεσία και υπάρχει και το θέμα του due diligence σε δέωσα επιμέλεια παραδείγματος στην αλυσίδα παραγωγής κάποιων επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο το ανέφερα ε, στην παρέμβασή μου ότι πρέπει δηλαδή στο εταιρικό δίκαιο, παραδείγματο χάρη, να μπορούν οι επιχειρήσει να ορίζουν μακροπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου κλιματικού στόχου, αλλά και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μπορούμε να επαληθεύουμε του στόχου αυτού και να βλέπουμε κατά πόσον εκεί συμμετέχει όλη η αλυσίδα παραγωγή. Τώρα, χρειάζεται αυτό να είναι ε, θέμα νομική υποχρέωση. Ε, θα σημειώσω την πρόταση και κατά πάσα πιθανότητα γιατί ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει, κατά πάσα πιθανότητα θα το συστήσουμε μαζί για να δούμε ποια είναι τα βήματα από εκεί και πέρα. Ε, επιβεβαιώνω όμως αυτό που είπα στην αρχή τη παρέμβαση. Σίγουρα δεν αρκούν ε, οι ε, εθελοντικές διαδικασίες και ο θελής προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. κύριε Ομπρή, άλλο ένα λεπτό στη διάθεσή σα. για να διευκρινίσω, δεν θέλουμε να ζητήσουμε από τι επιχειρήσει, αλλά θέλουμε να είναι δυνατόν να προσφέρουν στη δικαιοσύνη τα θύματα που δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Στη γραπτή σα απάντηση που τη μελέτησα με μεγάλη προσοχή λέτε ότι πριν υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα πρέπει να αξιολογούνται τα συμβάντα και ο αναλογικό χαρακτήρα όλων των μέτρων ε, για το θεμητό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Εμένα τι με ανησυχεί. Στο Βέλγιο στηρίζεται... Ε, έναν ε, νόμο που ουσιαστικά επιτρέπει στις επιχειρήσεις ε, να μην ε, πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Πείτε το ξεκάθαρα λοιπόν, ως αρμόδιος για τη δικαιοσύνη επίτροπος, η ελεύθερη αγορά θεωρείται ότι τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες τους τοποθετούν εκτός δικαίου, γιατί περί αυτού πρόκειται σήμερα. Εμείς θέλουμε να πάψει το φαινόμενο της μαρισίας των πολιεθνικών. Θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει να μπαίνει πάνω από το κοινικό συμφέρον, το συμφέρον των επιχειρήσεων. Να απαντήσετε. Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρη, κυρία Ομπρή. Φυσικά και δεν θεωρώ ότι όπω και οποιοδήποτε άλλο θα έπρεπε η επιχείρηση να είναι εκτό δικαίου. Φυσικά και πρέπει να είναι εντό κράτου δικαίου και επιχειρήσει, όπω και οποιοδήποτε άλλο παρά. Επειδή μιλήσετε για αναλογικό χαρακτήρα, φυσικά και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με τα μέτρα που λαμβάνουμε, όπω απέναντι στου μικρομεσαίε επιχειρήσει, μεγάλε επιχειρήσει, στου πολίτε. Και το είπα ξεκάθαρα. Είδα τα τελευταία χρόνια, ιδίω στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, κάποιε δεσμεύσει και οθελεί ε, εθελοντικές. Δεν αρκούν αυτά και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Μέχρι πού όμως θα φτάσουμε, αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Είπα και επαναλαμβάνω ότι έχουμε και την ε, ίδια την επιχείρηση που θα πρέπει να κοινοποιεί πληροφορίες ό,τι αφορά το κοινωνικό συμφέρον ε, και δεν είναι μόνο βράχη πρόθεσμο, αλλά θα είναι μέσο και μάκρο πρόθεσμο. Θα πρέπει να αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όταν μιλάτε για τα μέσα που θα έχουν ε, οι δικαστικές αρχές αλλά και οι ελεγκτικές αρχές, ναι, πράγματι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι αρχές αυτές στις πληροφορίες ώστε να μπορούν να εγγυηθούν τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι και στις πολυεθνικές. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς αυτό. Γιατί μου είπατε αν θεωρώ ότι πρέπει να είναι εκτός ε, κράτους δικαίου επιχείρηση. Όχι, δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ε, ερωτήσεων με τους ε, συντονιστές και εκπροσώπους των κρατών μελών, των, σύγχρονων των πολιτικών ομάδων. Και τώρα θα προεδρεύσει η κυρία Νέτσιγκερ για τον επόμενο γύρο της συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτος που θα θέσει ερώτηση θα είναι ο κύριος Εμίλ Ραντεφ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ρέιντερς, στις απαντήσεις σας στις γραπτές ερωτήσεις της Γιούρη είπατε ότι χρειαζόμαστε συντονισμένη προσέγγιση ώστε να οικοδομήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δικαστικά συστήματα. Ε, στο ψήφισμα της 4ης ε, Ιουλίου το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για κοινά ελάχιστα πρότυπα ε, για τις αστικές διαδικασίες. Ως εισηγητής του θέματος αυτού πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη ανάμεσα στα συστήματά μας. Έχετε εσεί σκοπό να υποβάλλετε μια τέτοια νομοθετική πρόταση και εάν ναι, πότε μπορούμε να περιμένουμε μια τέτοια πρόταση. Δεύτερη ερώτηση. Εάν ε, διοριστείτε επίτροπος ε, δικαιοσύνη, θα προτείνετε ευρωπαϊκή στρατηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον κύριο Ράντεφ. Ε, ναι, είναι η απάντηση και σε ποια προθεσμία ε, σίγουρα από κοινού θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εργαστούμε και υπενθυμίσατε ότι αυτή η πρόταση έγινε το 2017 για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο πρώτα και μετά να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο. Το έχω πει και σε μια γραπτή μου απάντηση. Έχω έτσι μια μικρή εμπειρία από το Συμβούλιο. Ε, σε 41 διαδοχικές ε, προεδρίες ε, είχα συμμετοχή και πραγματικά θα πρέπει να αποφύγουμε εμπλοκές και αδιέξοδα. Για τα θέματα αστικού δικαίου ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ μεγάλες επιφυλάξεις και δισταγμοί. Από κοινού θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε εδώ πρώτα να αποσπάσουμε πλειοψηφία ό,τι αφορά τους προσανατολισμούς, στις γενικές κατευθύνσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι αντίστοιχο με το δικαίωμα πρωτοβουλία που θέλει να αναγνωρίσει τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο η, πρόεδρος, ε, η νέα πρόεδρος Κομισιόν. Σίγουρα, δυνάμει και του άρθρου 225 και στη βάση καλή συνεργασία και συνεννόηση μπορούμε να δεχτούμε τέτοιε προτάσει από το Κοινοβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, υπάρχει πρωτοβουλία ε, στο πλαίσιο του προγράμματο εργασία που είναι η ε, λειτουργία του, Ευρωπαϊκού, του, της, του Γραφείου Ευρωπαϊκή Αγγελία, που θα πρέπει να αναλάβει έντονε πρωτοβουλίε σε αυτό το θέμα. Στα τέλη του 2020 θα πρέπει να μπορεί να είναι επιχειρησιακό αυτό το γραφείο. Οπότε για πρώτη φορά θα μπορούμε να γίνονται έρευνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να γίνονται και ε, διώξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά αυτό δεν μα εμποδίζει από το να προσπαθήσουμε να, όπω είπε και η κυρία Κάνκο, να έχουμε μια καλύτερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δικαστικών συστημάτων, ώστε να είναι πιο ε, αποτελεσματική δίωξη ε, σε θέματα οικονομικού ή άλλου οργανωμένου έγκληματο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και φυσικά θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση αυτή. Αλλά από ευρωπαϊκή πλευρά πιστεύω ότι ένα πρώτο σημαντικό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παρακαλώ κύριε Ράντεφ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Η επόμενη ερώτησή μου είναι τι άλλα μέτρα προβλέπετε για να βελτιώσετε την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και να βελτιώσετε την δικαστική συνεργασία ώστε τα δικαστικά μας συστήματα να μπορέσουν να υποφεληθούν από νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Και με τον τρόπο αυτό να προωθηθεί και το εμπόριο. Κύριε Ράντεφ, να σας πενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη φυσικά και επιθυμώ η πρόσβαση αυτή να ε, συνοδεύεται από την προσφυγή στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, σχετίζεται με το κράτος δικαίου. Δηλαδή να είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αμερόληπτη σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό βέβαια ισχύει με τις διαδικασίες που έχουμε θέσει σε εφαρμογή εδώ και κάποιο καιρό για το κράτος δικαίου. Και θέλουμε να ενισχύσουμε την πτυχή ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ε, στο πίνακα επιδόσεων, σε αυτό το scoreboard που θα παρουσιάσουμε για τη δικαιοσύνη. Τώρα, υπάρχει ε, και η ανάγκη να πρικοδοτήσουμε ε, το πρόγραμμα δικαιοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ορισμένα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε κάποια δικαστικά συστήματα μηχανισμοί που επιτρέπουν την, ε, πρόσβαση, την καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ίσως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πλησιώσει τη διαδικασία αυτή, ιδίω για τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού υπάρχουν ομάδες πληθυσμού, το έχω δει στο Βέλγιο, έχουμε μηχανισμούς ενεργού υποστήριξη για να υπάρχει μια πιο άμεση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά του, για τι πρακτικέ τη βέλτιστε και όποτε χρειάζεται να παρέχουμε ενεργό υποστήριξη. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη ε, και η ΓΑΜΑ Δικαιοσύνη μπορεί να δώσει κάποια κονδύλια σε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να μα δώσει τη λύση. Thank you. The next question... Σας ευχαριστώ πολύ. Η Καταρίνα Πάλη, από την ομάδα SND και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρέντερ, τον τελευταίο καιρό είδαμε να δίνετε προτεραιότητα στην διαδικασία του άρθρου 7 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δεν κάνω λάθος, στις απαντήσεις σας δεν αναφέρεται το άρθρο 7 ούτε μία φορά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτό ότι θα χειριστείτε διαφορετικά την εφαρμογή του από ότι στην προηγούμενη θητεία, από ότι από τον Φραντ Τίμερμανς, ε, λιγότερο αυστηρά ενδεχομένως. Τι θα κάνετε όσον αφορά τις διαδικασίες του άρθρου 7. Κύριε Παλίνα, είμαι απόλυτα σαφής θέλω να προχωρήσω σε τέτοιες διαδικασίες, όχι μόνο στις συγκεκριμένε υποθέσεις που έχουμε, αλλά και σε άλλες υποθέσεις. Γνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχουν άλλα προβλήματα σε άλλα κράτη-μέλη. Εάν χρειάζεται, θα πρέπει να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε από τον κύριο Τίμερμαν. Έχω δει μια εξαιρετική έκθεση, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από το Συμβούλιο της Ευρώπης Η έκθεση αυτή δείχνει ότι ήταν απαραίτητη η εκκίνηση της διαδικασίας. Αποτελεί λοιπόν μέρος της εργαλειοθήκης μας, αλλά προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε και άλλα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας, να είναι ο μηχανισμός και η ετήσια έκθεση, που προσπαθώ να εκπονήσω για την πρώτη χρονιά της ε, νέας θητείας, διότι ε, θα πρέπει να έχουμε μία σοβαρή παραβίαση του κράτους δικαίου. Θα πρέπει όμως να αποστέλλονται συστάσεις στα κράτη-μέλη και παρατηρήσεις χωρίς διακρίσεις. Εξεπλάγει που επί τόσα χρόνια ήταν δυνατόν να σχολιάζουμε την δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών, κάτι απαραίτητο, όχι όμως να σχολιάζουμε τις κοινέ μας αξίες και αυτό είναι σημαντικό στο Συμβούλιο με την αξιολόγηση ομοτήμων, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, έκθεση στο Κοινοβούλιο. Ε, θα πρέπει να γίνεται αυτό. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μου, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 7. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι όσον αφορά την Ουγγαρία, Ρώτησα στο Συμβούλιο, είναι θέση όμως και της παρούσας Επιτροπής να είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να εξηγήσει τη θέση του, διότι η διαδικασία ξεκινάει από το Κοινοβούλιο. Είπα όμως στην πρώτη μου απάντηση ότι θα οργανώσουμε και διάλογο με όλα τα κράτη-μέλη για να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, ε, να προλάβουμε οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Παλή, και στη γραπτή σας απάντηση και σήμερα είπατε ότι όσοι να προστατεύονται τα δικαιώματα ε, των κατηγορουμένων σε ποινικέ διαδικασίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μέτρα θα λάβετε για να το πετύχετε αυτό. Επίσης, ε, τονίσατε την ανάγκη για ε, ενισχυμένη δικαστική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο είναι επαρκές για να έχουμε Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα χωρίς να υπονομεύεται το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα εάν οι εθνικοί εισαγγελείς ε, ε, αναγκαστούν να κάνουν πίσω ε, για τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρώτη μου ανησυχία, η πρώτη μου φροντίδα θα είναι να έχουμε σωστή εφαρμογή μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς ε, συνεργαστώ με τον ε, Ισαγγελέα και με όλους τους υπόλοιπους φορείς για να το πετύχω αυτό. Είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται να εργαστούμε πάνω και στα δύο στοιχεία που αναφέρετε. Καταρχάς πρέπει να γίνουν πολλά για να έχουμε καλύτερη προσέγγιση, να έχουμε μία κοινή σειρά ε, διαδικαστικών κανόνων. Έχουμε διαφορετικά συστήματα και θα πρέπει να εξετάσουμε τις διαφορές τους. αλλά πρέπει να υπάρχει απόλυτο σεβασμός ε, του κράτους ε, δικαίου, ε, κάτι που σχετίστηκε και με το άρθρο 7. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Από την άλλη, ίσως χρειαστεί να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ως πρώτο στοιχείο θέλουμε να συμπεριλάβουμε και την τρομοκρατία. Εάν όμως διασυνοριακά αντιμετωπίζουμε την ε, τρομοκρατία και όχι μόνο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα χρειαστεί περισσότερος ε, προϋπολογισμός, θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι, διότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τρομοκρατία. Θέλουμε όμως ένα κοινό όραμα όσον αφορά τους διαδικουστικούς κανόνες και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Κάριν Μέλκιορ από την ομάδα Ρενιού. Κύριε Επίτροπε, ε, μπορείτε να απαντάτε κατευθείαν, δεν χρειάζεται να περιμένετε να σας δώσω εγώ το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναφερθώ στο θέμα της επίλυσης διαφορών σε πλατφόρμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ορίσει τους δικούς της κανόνες με ψηφιοποίηση των ε, πάντων από τις αγορές μέχρι τον δημοκρατικό διάλογο, οι Ευρωπαίοι πολίτες όλο και συχνότερα αναγκάζονται να επιλύουν διαφορές ε, εντό τη πλατφόρμα. Είναι δίκαιο όταν έχουμε μία διαμάχη με το eBay ή το YouTube, η ίδια η πλατφόρμα να επιλύει την διαμάχη. Επιπλέον, συχνά οι εταιρείε αυτέ βασίζονται σε χώρε εκτό Ένωση με περιορισμένη πρόσβαση. Η εξοδικαστική επίλυση διαφορών είναι σημαντικό τμήμα του συστήματο δικαιοσύνη. Βλέπουμε όμω μια ιδιωτικοποίηση μεγάλου τμήματος του συστήματος αυτού. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα καταναλωτών και πολιτών. Η Κομισιόν θα φτιάξει ένα ευρωπαϊκό υπόδειγμα επίλυσης διαφορών με πλατφόρμες και με βάση τον ανεξάρτητο διαμεσολαβητή που ήδη υπάρχει σε διάφορα κράτη-μέλη και με βάση άλλα στήματα που υπάρχουν στα συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα, κυρία Μελχιόρ, συμφωνώ μαζί σας πως υπάρχει ένα πρόβλημα με τις διάφορες ε, πλατφόρμες που έχουν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μια διαδικτυακή πλατφόρμα στοχεύει τον καταναλωτή εντός της Ένωσης, οπωσδήποτε ο Ευρωπαίος ε, καταναλωτής έχει τα ευρωπαϊκά του δικαιώματα. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Πρέπει να φροντίσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Και ακόμα και αν μια πλατφόρμα έχει έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι σαφές. Το δεύτερο στοιχείο έχει ξεκαθαρίσει ε, τι σημαίνει στόχευση και μια χώρα δηλαδή να στοχεύεται μόνο υπάρχει δυνατότητα αντίδραση και μπορούν όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη να έχουν την δυνατότητα να έχουν μια εξοδικαστική επίλυση ε, αλλά υπάρχουν 460 φορείς εξοδικαστικής επίλυσης ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε υπάρχει σχετική οδηγία την οποία πρέπει να δούμε. Αλλά γεγονό είναι ότι μπορούμε να πάμε παραπέρα. Γιατί είναι αδύνατο να πούμε ότι οι καταναλωτές πρέπει τελικά να καταλήξουν στο δικαστήριο για να λάβουν μια θετική απάντηση. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είπα ότι θα εργαστούμε τη δυνατότητα μια συλλογική προσφυγής και μια σχετική οδηγίας, οπότε μια πρώτη απάντηση θα ήταν η δυνατότητα να έχουν την δυνατότητα πολλοί καταναλωτές από κοινού να προσφύγουν. Από την άλλη, συμφωνώ ότι πρέπει να σκεφτούμε νέους ε, μηχανισμούς. Τώρα δεν θέλω να σα δώσω συγκεκριμένη απάντηση να πω διαμεσολαβητή ή κάτι άλλο, αλλά πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τα διαφορετικά είδη εναλλακτική επίλυση διαφορών εντό τη Ένωση και ίσω να δώσουμε και περισσότερε πληροφορίε γιατί υπάρχει έλλειψη πληροφοριών στου καταναλωτέ. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο και να προσφύγουν και ότι υπάρχουν και εσωτερικοί μηχανισμοί επίλυση διαφορών. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας και την ε, δέσμευσή σας για να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση του συστήματος δικαιοσύνης. Επίσης χάρηκα που είπατε ότι θα μειώσετε τον αριθμό των ανασφαλών προϊόντων στις διάφορες πλατφόρμες. Όμως οι πλατφόρμες αυτές δεν διανέμουν μόνο απτά αγαθά αλλά και ψηφιακό περιεχόμενο. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιες ασάφειες όσον αφορά την αστική ευθύνη κάτι το οποίο καταλήγει σε Αποκλήσει. Αυτό επηρεάζει ζητήματα όπω η ελευθερία έκφραση των Ευρωπαίων πολιτών στι διάφορε πλατφόρμερ στο διαδίκτυο, Καθώ ε, συχνά χρησιμοποιείται η αυτόματη λήψη αποφάσεων υπομορφή φίλτρων. Πώς θα διασφαλίσετε πως ε, θα διασφαλισετε πώ θα μπορουσε να υπάρχει η άμεση ή έμεση εντολή τα φίλτρα αυτά να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Να ήθελα να πω ότι βλέπετε ε, στην ε, δήλωση της Προεδρού υπάρχει η δέσμευση ότι τις πρώτες 100 μέρες θα εργαστεί για μια προσέγγιση για τον ψηφιακό κόσμο και είναι ακριβώς ε, κομμάτι αυτό της δουλειά πολλών επιτρόπων και οπωσδήποτε και σε συνεργασία εγώ με τον εκτελεστικό πρόεδρο θα καταθέσω μια πρόταση για την δεοντολογική πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, μιλάμε για τον αλγόριθμο. Ε, πρώτα απ' όλα συλλέγουμε πληροφορίε. Ποια είναι η λογική ε, μια εφαρμογή. Δεύτερον, είναι δυνατόν για τον καταναλωτή να πει ότι δεν θέλω να με αντιμετωπίσει ένα αυτόματο σύστημα. Θέλω να έχω επαφή με άνθρωπο. Επίσης, είναι ε, σημαντικό οι αρχές, ε, οι εθνικές αρχές, οι φυσικές αρχές που έχουν τον έλεγχο, οι δικαστές δηλαδή, να μπορούν να αντιληφθούν το τι συμβαίνει. Γιατί αν δεν λάβει κάποιος ε, πληροφορίες, ε, δεν έχει δυνατότητα να δοκιμάσει μια εφαρμογή, δεν έχει δυνατότητα να αποφασίσει για την προστασία των καταναλωτών. Οπότε είμαι σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας τις πρώτες εβδομάδες για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να προστατεύσουμε μια τέτοια δεοντολογική και ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να περιμένουμε να υπάρξει μια αυτορύθμιση, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία... Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Πέτερς κατόπιν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά είναι αυτό το οποίο είπατε μόλις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ε, είμαστε πεπισμένοι πως υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι και ε, παραδείγμα χάρη η ασφάλεια του ε, αυτόνομου αυτοκινήτου ή των αυτόνομων όπλων παραδείγματο χάρη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει για την ώρα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και αυτό έχει κάποιους κινδύνους, ε, παραδείγματο χάρη ε, συστήματα που δεν ρυθμίζονται, που καθορίζουν όπως είπατε διάφορα δικαιώματα κτλ. Και από την άλλη τα κράτη-μέλη ε, θα αναπτύξουν την δική τους ρύθμιση στον τομέα αυτό. Είπατε λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρα μία αποστολή δική σας μαζί με την συνάδελφη την κυρία Βέσταχερ. Συγκεκριμένα λοιπόν αν μπορείτε να μου απαντήσετε ποιο χρονοδιάγραμμα βλέπετε ή θα είναι κλαδική ή οριζόντια η αντιμετώπιση. Πώς βλέπετε το νομικό πλαίσιο. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι να βελτιωθεί η πρόσβασή μας στα μεγάλα δεδομένα των μεγάλων επιχειρήσεων για να μπορέσουμε, όπως είπα, να επιτελέσουμε ένα ρόλο προστασίας. Και τέλος, υπάρχει ένα στοιχείο ελέγχου από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πέτερς. Σας είπα ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε τις πρώτες 100 μέρες να προχωρήσουμε σε ένα νέο πλαίσιο μιας τέτοιας ε, ε, εξέλιξης καθώς έχουμε έναν εξυγχρονισμό στην κοινωνία μας και υπάρχει όπως είπαμε ιδεολογική πτυχή ε, θα το κάνουμε, είναι σαφές, είναι ξεκάθαρο. Αναφέρθηκαν και κάποια παραδείγματα από την κυρία Μελχιόρ. Μετά τις πρώτες 100 μέρες, αφού γίνει μια κίνηση αρχής, θα έχουμε ένα οριζόντιο πλαίσιο και μετά βεβαίως θα περάσουμε στα κλαδικά στοιχεία. Ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη τις μεταφορές ή ό,τι αφορά την υγεία και διάφορα άλλα σημεία γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν ε, πιο εξειδικευμένα μέτρα. Αλλά το θέμα εδώ πέρα ε, στο πρόβλημα αυτό είναι ακριβώς η ευθύνη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα με ένα αυτόνομο αυτοκίνητο. Πού βρίσκεται, ξέρω εγώ, στους δρόμους των Βρυξελών. Γίνεται ένα τροχαίο. Ποιος είναι υπεύθυνο. Ο ιδιοκτήτης. Μπορεί να μην έκανε τίποτα αυτός ο κατασκευαστής ίσως. Αλλά και κάποιοι, ίσως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με νέες εφαρμογές, με νέες ε, τεχνολογίες επηρέασαν ε, το αυτοκίνητο. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε ε, πώς θα εξελιχθεί η νομοθεσία μας. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποια οδηγία, αλλά για την ευθύνη θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι δυνατόν να υπάρξει μια ταυτοποίηση της πραγματικής ευθύνης ενός στοιχείου σε μια αλυσίδα. Σας ευχαριστώ για την απάντηση και μια δεύτερη ερώτηση είναι ότι κάποιες αναλύσεις λένε ότι 70% των οικονομικών πλέον εκτιμάτων της επόμενης της οικονομικής ανάπτυξης ουσιαστικά της επόμενης δεκαετίας θα είναι σε ΙΠΑ και Κίνα τι ε, μπορούμε να κάνουμε επ' αυτού και ε, ποιοι είναι οι λόγοι τελικά για τους οποίους τόσο μεγάλο ποσοστό 70% θα πάνε στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα. Ε, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το ορίσουμε επακριβώς ένα ποσοστό. Κοιτάξτε, πρέπει να πάμε προς περισσότερη καινοτομία. Κάποτε θυμάμαι Ήμασταν σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισαβόνα πριν από 20 χρόνια και λέγαμε τότε σε 10 χρόνια θα είμαστε οι πρώτοι. Ε, εντάξει δεν τα καταφέραμε ακριβώς. Και μετά είχαμε το επόμενο έργα που λεγόταν Ευρώπη 2020. Σχεδόν τελείωσε και αυτό. Και πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε την καινοτομία, startups και τα λοιπά, επιχειρήσεις. Αλλά και με κάποιες προδιαγραφές για μια σωστή προσέγγιση με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων κτλ. Αυτό το βλέπετε παραδείγματο χάρη με την προστασία των δεδομένων. Με την ε, πάρα πολύ ισχυρή δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο και τώρα βλέπετε ότι έχει υπάρξει μια εξέλιξη σχετική στις ΗΠΑ. Εντάξει δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο α, έχουμε εμείς, αλλά υπάρχει μια πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε στην εξέλιξη μιας τέτοιας ε, τάσης πρέπει να σκεφτούμε την πραγματική συνεργασία μεταξύ καινοτομίας και υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εκεί πέρα νομίζω ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με, άλλους, ε, με άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βάουτερς τώρα. Ja, ehm, Καλώς ήρθατε κύριε Reinders. Έχω μια ερώτηση. Εδώ είμαι για την υποδηλασία που μάλλον όμως δεν είναι στη, στο χαρτοφυλάκιο σας αλλά ουσιαστικά θα στραφώ στις συλλογικές προσφυγές, συλλογική νομή προστασία. Είχαμε κάποια σκάνδαλα ε, τα τελευταία χρόνια με την Ryanair για παράδειγμα, με το Dieselgate, ε, με τα ε, μασχεύματα, μάλλον τα εφητεύματα μαστού ε, και το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολίτες που θέλουν να ε, ασκήσουν συλλογικά ε, μέσα, ένδικα μέσα. Ε, έρχομαι στην ποδηλασία, έρχομαι το ποδηλατό μου κάποιες φορές ε, στο κοινοβούλιο και όταν περιμένω στο φανάρι ε, αναπνέω τα καυσαέρια, είμαι σίγουρη, από πολλά ελαττωματικά οχήματα και όχι μόνο, αλλά και πολλοί άλλοι ποδηλάτες. Η ερώτηση μου λοιπόν εξή. γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αν εγώ έχω ένα Volkswagen, γιατί να μην μπορώ μαζί με τους άλλους γιατί να μπορώ μάλλον να ε, προσφύγω κατά της Volkswagen και να μην μπορώ να το κάνω αν αναπνέω τα καυσαέρια των αυτοκινήτων αυτών ως ποδηλάτης. Θα έπρεπε και οι ποδηλάτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε βάρος τέτοιων εταιριών, όπως η Volkswagen για παράδειγμα. Απάντηση, για να είμαι πολύ συγκεκριμένο, ε, κύριε Βόλτερς. Θέλω να πω ότι φυσικά πρώτα πρέπει να εγκριθεί η νέα οδηγία για να μπορεί να υπάρχουν ε, αυτά τα συλλογικά ενδικά μέσα και ελπίζουμε τον Νοέμβριο να έχουμε τη θέση του Συμβουλίου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα δηλαδή μέχρι τώρα. Εγώ πάντως συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει διαπιστευμένη ε, παράγοντες που θα μπορούν να πηγαίνουν. Αν ξεκινήσει αυτό θα μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο μπορούν και για άλλους λόγους να οργανώνονται τέτοιε διαδικασίες, όχι μόνο για τους καταναλωτές, για παράδειγμα. για τον αέρα των Βρυξελών που μπορεί να είναι μολυσμένος, αλλά παραδείγματο χάρη για το περιβάλλον και άλλους. Εγώ είμαι υπεύθυνο για την προστασία των καταναλωτών, εφόσον επιβεβαιωθώ. Ελπίζω λοιπόν το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο να έχουμε τη θέση του Συμβουλίου. για την οδηγία που θα μας επιτρέψει να έχουμε αυτή τη συλλογική ένωμη προστασία. Και αυτό θα είναι ένα παράδειγμα, ίσως. Δηλαδή ότι μπορούμε να δώσουμε δικαιώματα στους πολίτες οποιαδήποτε περίσταση. Θα μπορούσα λοιπόν να συζητήσω και με τους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι. Για το περιβάλλον, για παράδειγμα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να είμαστε ηγέτες ε, μετά από τη Συμφωνία των Παρισίων κτλ. Άρα, μετά την προστασία των καταναλωτών, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προστατεύσουμε τους πολίτες γενικώς όταν υπάρχουν παραβιάσεις στον τομέα αυτό. Και με τους άλλους επιτρόπους και με το κοινοβούλιο θα συνεργαστώ. Η οδηγία αυτή για τις ε, δράσεις αντιπροσώπευσης ε, θα στείλει ένα μήνυμα ότι μπορεί να υπάρξει λογική προσφυγή σε κάποιες περιπτώσεις προς των καταναλωτών και όχι μόνο από τους καταναλωτές. Σα Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να αναθυμίσω ή να ανησυχήσω. Και τα δύο είναι δυνατά, διότι είπατε κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Έπασε πτώση, θα το δω αισιόδοξα. Μπορείτε λοιπόν να δεσμευτείτε ότι θα κάνετε ε, ό,τι μπορείτε για να ξεμπλοκάρει το θέμα των συλλογικών προσφυγών στο Συμβούλιο και πώς θα το κάνετε αυτό και δεύτερον δεσμεύεστε να εξετάσετε αυτό που είπα ακριβώς πριν, να διευρυνθεί η οδηγία αυτή ώστε και άλλοι πολίτες που ανησυχούν να μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν. Ε, συγγνώμη, θα επαναλάβω, διότι ήμουν πολύ σαφής. Θέλω συμφωνία πάνω σε θέση του Συμβουλίου και αν αυτό είναι δυνατόν τότε τον Νοέμβριο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα χρησιμοποιήσω όλη μου την επιρροή και τις επαφές μου για να το πετύχω αυτό, αλλά γνωρίζετε ότι είναι δύσκολο θέμα. Ίσως θα καταφέρουμε τον Νοέμβριο και αν ναι τότε θα προχωρήσουμε με την οδηγία. Από την άλλη είπα ότι θα συνεργαστώ και με άλλους επιτρόπους ε, ε, αλλά και με το ε, κοινοβούλιο για να δούμε αν μπορέσουμε να διευρύνουμε τη δυνατότητα για συλλογικές προσφυγές και σε άλλους τομείς. Στέλνουμε σαφές μήνυμα και είναι δύσκολο να εξηγήσουμε ότι θέλουμε να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε διάφορους τομείς ε, χωρίς να λάβουμε ε, και πρωτοβουλίες. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι θα εργαστώ πάνω στο θέμα αυτό. Το είπα ήδη στην πρώτη μου απάντηση, σας το επιβεβαιώνω στη δεύτερη μου απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Χαουτάλα από τους Πρασίμουνους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Οριστέντα Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Η ερώτησή μου αφορά μια σημαντική πτυχή του κρατούς δικαίου. Όχι μόνο ο δικαστικός τομέας, αλλά και η κοινωνία των πολιτών ε, ε, δέχεται απειλές σε, σε πολλά θέματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Πώς θα προστατεύσετε ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών ε, που απειλούνται. Ένα πρόσφατο παράδειγμα θα ε, αναφέρω όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, ατόμων ΛΟΑΤΚΙ τα δικαιώματα αυτά απειλούνται. Είδαμε πρόσφατα επιθέσεις στην Πολωνία. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πώς θα προστατεύσετε την κοινωνία των πολιτών ε, και τα δικαιώματα των πολιτών. Σας ευχαριστώ κυρία Χαουτάλα για την ερώτησή σας. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση, διαδικασίες του άρθρου 7 για παραβίαση του κράτους δικαίου. Ε, πώς μπορούμε να είμαστε ε, πιο αποτελεσματικοί επιτόπου, στηρίζοντας τους διάφορους παράγοντες επιτόπου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να, γίνουν αυτό, ε, να γίνει αυτό. Και πολύ χαίρομαι που η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει να διατηρήσει τα ίδια επίπεδα χρηματοδότησης στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι δυνατόν όμως να στηρίξουμε και διάφορους παράγοντες ε, της κοινωνίας των πολιτών μέσω της χρηματοδότησης. Αυτός είναι ένας τρόπος. Άλλος τρόπος ε, είναι με την κατάρτιση ανθρώπων ε, και να συμβάλλουμε με επιρογνωμοσύνη από επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχουμε και αυτή την δυνατότητα. Θα είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις βασικές δύσκολες περιπτώσεις. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στον μηχανισμό που έχουμε με την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου και την επιλογή των προγραμμάτων που στηρίζουμε από την κοινωνία των πολιτών για να υπερασπιστούμε επιτόπου τα άτομα αυτά. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ και πολλά χρόνια ε, και ως Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου ε, ε, έχω ασχοληθεί με την προστασία των μειονοτήτων με τον τρόπο αυτό. Αυτή φυσικά είναι μία από τις ανησυχίες μας, υπάρχουν και άλλες ευάλωτες ομάδες, θα πρέπει όμως να δραστηριοποιηθούμε επί τόπου και όχι μόνο με τις γενικές διαδικασίες που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας. Οι πόροι λοιπόν είναι πολύ σημαντικοί, οι οικονομικοί πόροι, και θα προσπαθήσω να υπερασπιστώ τις δυνατότητες που έχουμε χρηματοδοτώντας σε διάφορους παράγοντες επιτόπου. Και ε, αν υπάρχει αιρεσιμότητα ε, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, σε σχέση με το κράτος δικαίου, θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοια προγράμματα. Θα είναι κρίμα να σταματήσει η χρηματοδότηση στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προς την κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην απάντησή σας προς την συνάδελφο Walters αναφερθήκατε στη Συμφωνία του Παρισιού. Κάποια θέματα λοιπόν προκύπτουν τώρα όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ε, σε σχέση με, την, ε, με το μετριασμό του κλίματος ε, και ε, έχουμε μια υπόθεση, ε, ε, έχουμε μια προσφυγή για παραβίαση των δικαιωμάτων μια ομάδας που αγωνίζεται για το κλίμα. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό, τους ανθρώπους που αγωνίζονται για το κλίμα και την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Εάν δεσμευόμαστε για κάτι, θα πρέπει να επαληθεύουμε και το εφικτό αυτών των δεσμεύσεων. Είναι δυνατό αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Κοινοβούλιο, ε, για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει και οι πολίτες όμως να μπορούν να διαπιστώνουν την ε, εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας. Ε, στο δικό μου πιθανό χαρτοφυλάκιο θα συμπεριλάβουμε μία δράση για να υπάρχει δυνατότητα συλλογική προσφυγή για καταναλωτέ. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα. Γιατί λοιπόν να μην σκεφτούμε παρόμοια προσέγγιση για πολίτε σε άλλου τομεί. με την ίδια προστασία. Μπορεί να χρειάζονται επιστοποιημένοι οργανισμοί για να το κάνουν αυτό, ε, να υπάρχει σαφής διαφάνεια και που να έχουν την δυνατότητα αποφυγής σύγκρουση συμφερόντων, διότι δεν ε, θα ήθελα να έχουμε παρόμοιες ε, συλλογικές ε, προσφυγές με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σας διαβεβαιώ όμως ότι θα εργαστικό πάνω στο θέμα αυτό. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Λεμπρετόν από την ομάδα ID. Παρακαλώ. Κύριε Ρεντέρ, η προτεραιότητά σας είναι το κράτος δικαίου να είναι σεβαστό σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Δύο μέρες έχετε ουσιαστικά στη διάθεσή σας ο περιοδικός έλεγχος της κατάστασης σε κάθε κράτος. Λίγο ανησυχητικά αυτό το λέτε ετήσια διαδικασία ένταξη και έπειτα οι οικονομικές κυρώσεις, δεύτερο μέσο. Όλα αυτά δεν ε, επηρεάζουν ε, πολύ τα εσωτερικά ουσιαστικά των κρατών μελών. Δεν είναι μια υπερβολική ανάμειξη. Επίσης, το κράτος δικαίου με μια ε, έννοια κάπως ευρία λέτε ότι περιλαμβάνει υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια των αγώνων για την κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα δεν θα τα βάλετε μόνο με την Πολωνία και τον Κάρλ, αλλά και με τη Γαλλία. Έχουμε τα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία μιλούν για έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης ε, και ε, έχουμε και το δημόσιο κατήγορο. Τι μέσα έχετε. Έχετε την κυρία Γιούροβα και τον Έλληνα Επίτροπο που έχουν λίγο πολύ τις ίδιες με εσάς αρμοδιότητες, ισοσμό των αξιών και από την άλλη στο ΒΕΛ έχετε τρεις θέσεις. Είστε υπουργό Εξωτερικών, υπουργό Άμυνα ε, ε, και φορματέρο Αγιάλ. Είναι ένα χάντικα αυτό. Πώς θα το ξεπεράσετε. Απάντηση. Πράγματι, ε, φορματέρ Ρουαγιάλ είναι μια έννοια που δεν υπάρχει σε πολλά κράτη βασιλικός πληροφοριώτης, κάπως έτσι. Δεν υπάρχουν, στην Γαλλία τα ξέρετε τα πράγματα. Λοιπόν, για την κατάσταση του κράτου δικαίου. Τι προσπαθούμε με αυτό το μηχανισμό να πετύχουμε. Είναι κάτι που το ζητάει το Κοινοβούλιο από τον Οκτώβριο του 2016 και το ζητώ και εγώ αρκετά χρόνια στο Συμβούλιο με την, ε, το αίτημα για την εξόριξη από μοντίμους. Είναι να μπορούμε να εκτιμούμε χωρίς διακρίσεις την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Το πώς θα γίνει εξαρτάται λίγο και από τα δημοσιονομικά. Υπάρχει ανάλυση, υπάρχουν συστάσει των οικονομικών κριτήριων τη Ένωσης. Σε επίπεδο Συμβουλίου και Κομισιών. Θέλουμε να μην υπάρχουν διακρίσεις, αλλά αν έχουμε σε κάποιο κράτος μέλος πρόβλημα, να λαμβάνουμε περισσότερη δράση. Αν δει κανεί το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, θα υπάρξουν συστάσεις και κριτικές. Ε, θέλουμε να έχουμε διάλογο ε, χωρίς διακρίσεις και θέλουμε να δράσουμε προληπτικά για να μην αναπτυχθούν καταστάσεις που μπορούσαν να δείξουν σε πραγματικές παραβιάσεις. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν θα πρέπει να δεχθούν να μιλήσουν για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις αξίες που είναι στο κέντρο του ευρωπαϊκού Οικοδομήματο. Όλοι μιλάμε για ένα οικοδόμημα που εδράζεται σε αξίε, Δεν, δεν ε, έχει σημασία να δούμε ότι πράγματι αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο των αξιών αυτών με τον ίδιο τρόπο και ότι μέσω εθνικών συμπεριφορών και νομοθεσιών εφαρμόζουμε σωστά του κανόνε του κράτου δικαίου. Και αυτό θα κάνουμε. Τώρα αν αυτό πάει πολύ μακριά, κοινωνική δικαιοσύνη εγώ νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδόμηματος. Φαίνεται προφανέ λοιπόν να ασχοληθούμε για να παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ένωση στον τομέα αυτό. Αυτό που θα ήθελα και το έχω ξαναπεί είναι να εργαστούμε από κοινού. Η Κομισιόν, μίλησα με την κυρία Γιούροβα, θα κάνει την έκθεση για το χάρτη των δικαιωμάτων, θα έχουμε ε, για τη δημοκρατία επίσης άλλα σε τέτοιες εκθέσεις. Ε, θέλω λοιπόν να έχουμε μία συζήτηση σε βάθος και να γίνει διοργανική, γιατί σίγουρα έχει τη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Όμως, εγώ επιμένω και ε, επαναλαμβάνω ότι έχετε τρεις ε, θέσεις. Δεν είναι αυτό το μοντέλο που εγώ θα ήθελα να δω για... σε σχέση με το κράτος δικαίου. Πριν κοπεί το ρεύμα, είχατε πει σωστά ότι ε, δεν θέλετε τόσο τις κυρώσεις ε, και προτιμάτε την πρόληψη. Με ανησυχεί όμως κάτι που είπατε, είπατε αιρεσιμότητα μεταξύ του πι δέλτα πι και του κράτους δικαίου. Και καταγγείλατε την εθνικιστική ρητορική. Είπατε ότι υπάρχουν κράτη που θέλουν να κυριαρχήσουν και όχι να συνεργαστούν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρω σε ποιο κράτος αναφέρεστε συγκεκριμένα. Όλα αυτά δείχνουν ε, μία ένωση που θέλετε να είναι ε, τελικά ομόσπονδη και την ελευθερία του κάθε ευρωπαϊκού έθνους πώς την αντιλαμβάνεστε. Ο κύριος ε, Ράιντες. Να σας καθησυχάσω ότι τις, τα τρέξω με στο θα τα εγκαταλείψω εφόσον επιβεβαιωθώ ως Επίτροπος. Δεύτερον, όταν μίλαγα για έθνη, νομίζω ότι ε, μιλούσα για κράτη εκτός Ένωσης που μονομερός δρούν και όλο και λιγότερο συμμετέχουν στο πολυμερές σύστημα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε ε, ποια είναι αυτά τα έθνη. Η Ευρώπη είναι ένα χώρος πολυμερούς δράσης ε, από τους πλέον εξέχοντες. Το ευρωπαϊκό οικοδόμα εδράζεται στη βούληση, στη θέληση των κρατών μελών να προχωρήσουν λίγο, λιγότερο ή περισσότερο στη συνεργασία τους. Φυσικά και αφήνω χώρο και περιθώρια ε, στα κράτη να ασκήσουν τις πολιτικές τους. Όμως κάθε φορά που θα θεωρούμε ότι υπάρχει μια προστιθέμενη αξία με μια κοινή δράση και ιδίως απέναντι σε διεθνείς ε, ε η απόφαση ίσως θα πρέπει να λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη ή τις κυρώσεις. Αν έχουμε την αιτήσια έκθεση και αυτό μηχανισμό, φυσικά και θα δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και δεν θα μείνουμε μόνο στη λογική τη επιβολή κυρώσεων. Το είδαμε τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα θα συνεχίσουμε, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσουμε το σκέλο αυτό και με την πρόληψη. Ευχαριστώ. Σταν Κανέλη, να επόμενο από το ECR. Eh, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σύμφωνα με την Υπηρεσία για την Προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων, οι απώλειες ε, λόγω της ε, πειρατείας τομείς κλειδιά όπως ο ρουχισμός, φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα κτλ είναι γύρω στα 60 δισεκατομμύρια το χρόνο και στην Ιταλία υπολογίζεται ότι το ποσό ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος. Η εκτίμηση της υπηρεσίας αυτής λέει επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη χάνονται μέχρι και 468.000 θέσεις εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν θα ασχοληθείτε με την προστασία των ε, καταναλωτών και πώς θα μπορέσουν να κάνουν επιλογές ενημερωμένοι όσον αφορά το εάν αγοράζουν κλεψίτυπα προϊόντα και τι σκοπεύετε να κάνετε ακριβώς για να καταπολεμήσετε αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή για το ρόλο που μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε κατά τις παραποίησης Σίγουρα είναι μια εγκληματική δραστηριότητα η παραποίηση, οι ε, και οι τελωνικέ υπηρεσίε ε, πρώτα απ' όλα εργάζονται για να ανοιχνεύουν, εντοπίζουν ε, διασυνοριακή μεταφορά τέτοιων εμπορευμάτων και με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο για την οικονομία θα το συστήσουμε στο μέλλον το θέμα αυτό, αλλά σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη επιβάλλει σε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν κυρώσει σε όσου εμπλέκονται σε δραστηριότητε παραποίηση ή και πειρατεία. Στον τομέα τώρα της δικαιοσύνη, το Eurojust συγκεκριμένα θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών, ε, ιδίω ε, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με την πραγματική ιδιοκτησία. Εδώ σίγουρα πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση μας. Μάλιστα εκπονεί και μια έκθεση για τις προκλήσεις και για τις βέλτιστες πρακτικές από δικαστικής πλευράς για την αντιμετώπιση αυτού του είδους της εγκληματικότητας. Δηλαδή έχουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών. Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Πρώτα απ' όλα οι πλατφόρμες, οι ψηφιακές πλατφόρμες, αν μιλάμε για ε, διαδικτυακές πωλήσει, θα πρέπει να κάνουν πάντα δυνατό για να αποτρέπουν ε, τις ε, πωλήσει, αγοραπολισίες παράνομων προϊόντων όταν αυτά θα έχουν εντοπιστεί. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τις πλατφόρμες, γίνεται αυτό στο πλαίσιο ενός δικτύου ε, των αρχών προστασίας των καταναλωτών και μπορούμε να προχωρήσουμε από αυτού. Νομίζω ότι με στατιστικές και με δεδομένα τα οποία τώρα συλλέγουμε, θα μπορέσουμε να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό ο τομέα. Όπω είπατε και εσεί, θα έχουμε όλο και πιο στενή συνεργασία και με τη Eurojust. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προβλέπει ήδη την επιβολή κυρώσεων θα αναλύσουμε αν χρειάζεται να πάμε πιο πέρα. Γιατί προς το παρόν νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να ενισχυθεί πολύ είναι ο συντονισμός. Eh, Σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν ανέφερε μία αρχή. Ε, κάθε νομοθέτημα που θα έρχεται σημαίνει ότι θα καταργείται ένα άλλο. Λοιπόν, ε, ποια σκοπεύετε εσείς να καταργήσετε για τα νομοθετήματα τα οποία θα φέρετε, ειδικά όσον αφορά τη μηματική ιδιοκτησία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να υπερασπιστείτε την έρευνά τους, την δραστηριότητά τους ε, που με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα στην οικονομία Πρώτα απ' όλα να σας ομολογήσω ότι δεν έχω ε, κάνει ένα κατάλογο με τον νομοθετήματα που θα έπρεπε να αποσυρθούν ή να καταργηθούν ε, και στις γραπτές μου πατήσεις και στην εισαγωγική μου παρέμβαση είπα ότι θα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε, να αναθεωρήσουμε κάποια νομοθετήματα, κάποιε οδηγίες, ιδίως ότι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια που ήδη καταβάλλεται ώστε να περιοριστεί το διοικητικό άχθος να περιοριστούν τα διέξοδα και εμπλοκέ που σίγουρα βαρύν το έργο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νοφιών επιχειρήσεων που δεν έχουν τι ίδιε δυνατότητε, όπω οι μεγάλοι όμιλοι, ή οι πολυεθνικές μπορούν να, ανταποκριθούν πιο εύκολα στις υποχρεώσει που του επιβάλλουμε. Επίση, προστασία δεδομένων. Ακούω πολλέ φορέ κριτικέ για αυτό το γενικό κανονισμό σας δεδομένων. Όμως, ο κανονισμό αυτό περιλαμβάνει προστευμένους μηχανισμού για τις ΜΜΕ. Σε αυτό το πνεύμα πιο πολύ θέλω να εργαστώ. Δηλαδή, ή δυνατόν ορισμένα νομοθετήματα ε, να μην ε, περιλαμβάνουν αχρίαστες υποχρεώσεις που δυσκολεύουν το έργο των νεοφιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Πριν περάσω στον κύριο Αριμών, θα ήθελα να πω στους βουλευτές ότι έχουμε καθυστερήσει λίγο, οπότε σας παρακαλώ να περιοριστείτε απολύτως στο ένα λεπτό. Και πάντα καταφέρετε και σε λιγότερο από ένα λεπτό, ακόμη καλύτερα. Έχετε τον λόγο. Καλημέρα σας ε, και καλώς ήρθατε. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Θα ξέρετε οπωσδήποτε τον κανονισμό περί δικαιωμάτων ε, αεροπορικών επιβατών. Ε, πιθανώς γιατί τη γνωρίζουν πάρα πολλοί καταναλωτές στην Ευρώπη και είναι πάρα πολύ ευνόητος αυτός ο κανονισμός γιατί είναι ίδιος και στα 28 κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει όμως, ε, είχαμε κάνει μια πρόταση, να συμφωνήσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη σε μια συγκεκριμένη διάρκεια της εγγύησης των ε, καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Γιατί δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 10 άτομα, ούτε ο καταναλωτής να ανταποκριθεί σε 28 διαφορετικά κασότα. Αυτό μπορεί να το κάνουν μόνο μεγάλες εταιρείες. Θα, λοιπόν, θα πρέπει να είναι κάτι το απλό και ενιαίο. Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου πως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να είναι ευνόητοι και ίδιοι. Συμφωνείτε δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση των κανόνων σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο στόχος αυτός πρέπει να είναι, άρα συμφωνώ απόλυτα και η απάντηση μου είναι ναι για τη βούληση προς εναρμόνιση και αυτά που είπατε για τις εγγύησει. Ε, σίγουρα οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυτό το ρίσκο που είπατε όταν απευθύνονται σε διάφορους προμηθευτές. Καλό είναι να υπάρξει μέγιστη δυνατή εναρμόνιση τη προστασία των καταναλωτών. Αυτό έχει γίνει με πολλά κείμενα προσφάτω. Δηλαδή να έχουμε αυτή τη λογική τη προστασία με τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση. Φυσικά θα πρέπει να δούμε κατά περίπτωση τα πράγματα, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει, όχι τόσο στη δική, στο δικό σα παράδειγμα, θα πρέπει να επιτρέπουμε νιώτε σε κάποια κράτη-μέλη να ευθετήσουν ε, περισσότερα μέσα προστασία απέναντι, παραδείγματο χάρη σε βάλου καταναλωτέ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει υπόψη σε ορισμένου ε, τομεί. Αυτό το θέμα για τι αεροπορικέ εταιρείε, δικαιώματα επιβατών, πράγματι είναι πολύπλοκη κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή με την τόση σχέση ενό ταξιδιωτικού γραφείου. Ε, η κατάσταση βέβαια από ό,τι φαίνεται ε, όταν μιλάμε για 600.000 άτομα εξελίσσεται πολύ καλύτερα γιατί θα μπορούσε να υπάρχει ένα πλήρε χάο. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν πτωχεύσει μια αεροπορική εταιρεία. Νομίζω ότι και εκεί πρέπει να γίνει ε, κάποια δουλειά, ε, ώστε σε ευρωπαϊκή κλίμακα να υπάρχουν κάποια εγγυημένα δικαιώματα, ώστε το δυνατόν, επαναλαμβάνω, πιο εναρμονισμένα για του επιβάτε αν κάνουμε τη σύγκριση όχι με το τι έχει γίνει κατά παρελθόν, αλλά τώρα με την πτώχευση του στομακού, Για να πω με το όνομά του ποιο είναι αυτό, το, ποια είναι αυτή η εταιρεία που πτώχευσε. Και αύριο ξέρω ότι θα υπάρξουν ε, σχετικέ εργασίε σε σχέση με τι αεροπορικέ εταιρείε. Συμφωνώ όμω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εναρμόνιση προσέχοντα τι ομάδε ε, ομάδες των πιο ευάλωτων καταναλωτών και βλέποντας τα κράτη που θέλουν να προχωρήσουν σε μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας. Σα ευχαριστώ για την απάντηση. Θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα και θέλω να σα ρωτήσω εάν είστε διατεθειμένοι να κάνετε έναν έλεγχο σε όλους τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και να μας πείτε πού μπορεί να γίνει η πλήρης εναρμόνιση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. δεύτερη ερώτηση Σύμφωνα με την επιστολή ανάθεσης ε, καθηκόντων, ε, είστε υπεύθυνο για να αναπτύξετε μια στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είπατε στον συνάδελφο πριν ότι θα δείτε ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν, αλλά μπορείτε εδώ να μας πείτε ποια συγκεκριμένα μέτρα θεωρείτε εσείς ε, ότι θα διευκολύνουν την ζωή των μικρομισών επιχειρήσεων που δημιουργούν ε, το 90% σχεδόν των θέσεων εργασίας ε, στην Ευρώπη. Ε, συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις 10 ανθρώπων, όπως μου αρέσει συχνά να λέω. Πώς θα τους απλοποιήσετε τη ζωή να απαντήσω και στι δύο ερωτήσει. Πρώτη ερώτηση, απάντηση είναι ναι. Νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Σε σχέση όμω με την απάντηση που έδωσα στην πρώτη σα ερώτηση, όπου είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση, είναι μια εγγύηση αυτό που μπορούμε να δώσουμε στου καταναλωτέ. σω υπάρχουν κάποιε περιπτώσει όπου μια επαλήθευση θα δείξει ότι πρέπει να αφήσουμε κάποια περιθώρια σε όσα κράτη-μέλη θέλουν να πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να ε, κάνουμε. Τώρα, ε, σας μίλησα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αλλά υπάρχει η ψηφιοποίηση που ε, γίνεται όλο και ευρύτερη στην νομοθεσία που θα πρέπει να θετήσουμε από αυτού. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ περισσότερο τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχουν τον, τη θέση τους σε αυτή την ψηφιακή εποχή και όχι να επιβαρυνθούμε τους κανόνες που επιβάλλουμε. Αυτό γίνεται με το Γενικό Κανονισμό. Υπάρχουν ειδικοί στις διατάξεις της ΜΜΕ. Πρέπει να δώσουμε προσοχή λοιπόν στα μέτρα τα οποία θα λάβουμε όταν θα θέλουμε να ε, δούμε την νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως. Θα υιοθετήσουμε. Σας... Η ε, κυρία Παγάθα Ουρτουντούα είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είπατε κύριε Ρέιντερς ότι αλλάζει ο κόσμος ε, και υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση και σε ό,τι αφορά το ε, έγκλημα και την ατιμορρησία. Είπε η κυρία Γιώχανσον ότι θα πρέπει η αρχιτεκτονική της δικαστικής συνεργασίας να είναι έντιμη για να μην υπάρχουν κρασιμία και για να αντιμετωπιστούν οι νέες και αναδυόμενες απειλές. Το ίδιο ισχύει και στην δικαστική συνεργασία. Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσματική των δικαστικών αποφάσεων στον κοινό χώρο ελευθερία και δικαιοσύνη, να μην υπάρχουν καταχρήσει. Θέλουμε περισσότερε εγγυήσει και θέλουμε να προασπίσουμε τα νομικά δικαστικά ε, συστήματα και το κράτο δικαίου με το ευρωένταλμα. Δεν θα πρέπει αυτά τα σοβαρά εγκλήματα να είναι ατιμόρυτα. Υπάρχει νομίζω σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση των αξιόπινων πράξεων ε, περιθώριο βελτίωσης ε, για την προστασία των νομικών αγαθών και κυρίως το κράτος δικαίου και την δαφική ακαιρεότητα, το κράτο του νόμου. Νομίζω ότι τι με, είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι με το, με το ευρωένταλμα. Θα, θα γίνει αυτή η αναθεώρηση και η βελτίωση. Σας ευχαριστώ που επανέρχεστε στο ένταλμα. Ε, σύλληψης. Ε, η συνεργασία μεταξύ των δικαστικών συστημάτων είναι κάτι το οποίο γίνεται και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα τη Ένωση, το είπα, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ε, φορέα που θα κάνει έρευνε και θα κινεί διώξει και θα έχει και ευρύτερε αρμοδιότητες κατά πιθανότητα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα εγώ θα πω ότι είναι success story. Είναι μια επιτυχημένη προσέγγιση είχαμε εντάλματα που στο 50% έγιναν δεκτά και αυτό έχει μειώσει πάρα πολλές προθεσμίες ε, στις 16 ε, μέρες. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Και επειδή υπάρχουν αποφάσεις του δικαστηρίου, καμιά σαρανταριά, που μας δίνουν τη δυνατότητα πλέον να βελτιώσουμε ε, τις κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνουμε στα κράτη-μέλη, για να υπάρξει αυτή η ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας των διώξεων αφενός, γιατί όπως είπατε είναι σοβαρά τα εγκλήματα αυτά και το δικαίωμα της υπεράσπισης από την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή κάνει την αξιολόγηση της κατάστασης και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν σωστά Άρα, όπω ζητάτε, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, ότι εφαρμόζει σωστά τι ευρωπαϊκέ διατάξει. Και σε περίπτωση που δεν είναι προφανές ε, να κινηθεί η δικασία παραβάση σε βάρος αυτών των χωρών. Υπερθύμησα επίσης και κάτι άλλο. Αν από αυτή την αξιολόγηση αποδειχθεί ότι καλό είναι να γίνουν τροποποιήσει ε, στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, εγώ είμαι απολύτω ε, έτοιμο και διατεθειμένο να καταθέσω μια τέτοια πρόταση αναθεώρηση, βεβαίω στο πλαίσιο διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είναι υπέρ τη αναθεώρηση και την οποία μετά θα καταθέσω και στο Συμβούλιο. Πάντω, ναι, πράγματι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση ορισμένων σοβαρών εγκλημάτων, εξώπινων πράξεων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέιντερς για την δέσμευση. Για κάθε μία από τις βελτιώσεις και κάθε ένα από τα στοιχεία ε, για τη βελτίωση της οδηγίας σίγουρα ε, θα κάνουμε και εμείς ακούραστα τη δουλειά μας. Ε, στη δεύτερη ερώτηση θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι είπατε στις γραπτές απαντήσεις ότι θέλετε να εφαρμοστούν σωστά οι διατάξεις οδηγίας για τα ελάχιστες διατάξει ότι αυτά τα δικαιώματα στήριξη, προστασία των θυμάτων το 2012. Υπάρχουν πραγματικά ε, αυτές οι ανάγκες. Έχουμε θύματα που έχουν υποστεί φοβερά εγκλήματα, με, αφήνουν τραύματα και σίγουρα ε, σε αυτή την οδηγία καθορίζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αλλά μιλάμε για τα ελάχιστα. Καλά είναι τα λόγια, αλλά εμείς βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται αυτό το πλαίσιο από τα κράτη-μέλη το 2018 συγκεκριμένα, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ το 2017 ε, είχε αναθέσει τη διεξαγωγή έκθεση για να δούμε τι ε, λύματα υπάρχουν για την προστασία των θυμάτων σοβαρών εγκλημάτων. Χρειάζεται λοιπόν, κύριε Ρέιντερ, ένα επαναστάτη επίτροπο που δεν θα μείνει στα, ε, ε, στα απλά καλά λόγια, αλλά θα βοηθήσει τα θύματα. Θα είστε εσεί αυτό ο επίτροπο απάντηση. Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα πάνω σε δύο από αυτά που είπατε. Ναι, ότι πράγματι θα πρέπει να δούμε πραγματικά οι διατάξεις και οι δεσμεύσεις αν εφαρμόζονται. Ε, και ιδίως για τα θύματα της τρομοκρατίας, για παράδειγμα, γιατί δεν ήμασταν μόνο εδώ, σε Βρυξέλλες και σε πολλές άλλες πόλεις του κόσμου, χτύπησε η τρομοκρατία με πολλά θύματα και πρέπει να, εφαρμοσ να δούμε αν εφαρμόζονται σωστά ε, αυτά. Αλλά δεύτερη παρατήρηση εδώ. Δεν αφορά αυτό μόνο θύματα τρομοκρατίας. Ε, υπάρχουν ε, και άλλα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε την δυνατότητα πρόσβαση, ενημέρωση των θυμάτων, πλαισίωση των θυμάτων, υποστήριξή του. Υπάρχει ένα πιλωτικό σχέδιο για την τρομοκρατία αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαμε ίσω να το ε, διευρύνουμε, να περιλαμβάνει όλα τα ε, άλλα εγκλήματα. Είναι 41 οι συστάσεις της ε, έκθεσης που συνέταξε εκ μέρους του κυρίου Γιούνκερ, η Μιλκέτ, και πράγματι μπορούμε να τα μελετήσουμε όλα αυτά. Σα Σας ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση της κυρίας Βίντικαμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν ευγνώμων για την ειλικρίνεια του οριστέντα επίτροπου σχετικά με τα ε, προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει, σχετικά με διάφορες κατηγορίες. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως το εξή. Δεδομένου ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε πολύ σαφώς στην επιστολή ανάθεση καθηκόντων ότι δεν, μπορεί, δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την ακαιρεότητα και τη συμπεριφορά ε, επιτρόπων, ε, εξέτασε το ενδεχόμενο παρέτησή του μέχρι να λυθεί το θέμα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Thank uh, Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως ε, είπα στην εισαγωγή μου, ο εισαγγελέας είπε ότι δεν υπάρχει κατηγορία και γι' αυτό δεν παρετούμε. Ε, θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ε, και συνεχίζω να το κάνω αυτό ακούστηκαν νέες ε, κατηγορίες. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι εκατοντάδες ε, χιλιάδες αθώοι πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορούνται λανθασμένα και έχουν χάσει τη δουλειά τους ή δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για κάποιες θέσεις. Τι εικόνα θα έχουν αυτοί όταν οι ηγέτες ενός τεράστιου φορέα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διορίζει ανθρώπους που ε, δεν έχει αποδειχτεί ακόμα η αθότητά τους. Ε, υπάρχει βέβαια η αρχή ότι είναι κανείς αθώος μέχρι να αποδειχτεί ένοχος, υπάρχει όμως και ισότητα απέναντι στον νόμο. Ναι, πράγματι, ε, αλλά αυτό ισχύει για όλους ε, και για μένα. Και ε, στην πρώτη υπόθεση ο, ο δικαστής και ο εισαγγελέας ήταν σύμφωνοι. Εάν ξαναπροσφεύγουν η απάντηση παραμένει η ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χαλτζεράν από το S&D. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιο επιτροπέ. Εάν διοριστείτε ένα από τα καθήκοντά σας θα είναι να διασφαλίσετε ότι προστατεύονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή γενικώ και στην ε, τεχνητή νοημοσύνη ειδικώ. Αναφερθήκατε ήδη εν μέρη στο θέμα, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επεκταθείτε και έχω τις εξής ερωτήσεις. Πώς θα εγγυηθείτε την εγγύηση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης στις διαδικασίες συλλογής και εφαρμογής προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη πως έχουμε ήδη παραδείγματα αλγοριθμών που ρουφιανεύουν, ε, κάνουν λανθασμένες προβλέψεις κτλ. Δεύτερον, βλέπουμε ότι αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο και καμιά φορά χρησιμοποιούνται, ε, δημιουργούνται κιόλας για σκοπούς επιβολής του νόμου. Πώς ε, θα φροντίσετε να γίνονται σεβαστές ε, οι αρχές της αναλογικότητας και μία σύντομη ερώτηση, με ναι ή με ένα όχι. Θα φροντίσετε η με οχι θα φροντισετε η κομισιον να φροντίσει να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και στον τομέα επιβολής του νόμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη δεύτερη ερώτηση, η απάντηση είναι ναι. Δεν είναι ζήτημα το έχω πει αυτό και πολλές φορές ε, είναι το πρώτο στοιχείο του χαρτοφυλακίου με αν το αναλάβω να υπερασπιστώ τα ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επαναλαμβάνω και για την τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να πάμε προς καινοτομία, νέα προϊόντα κτλ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι να το κάνει αυτό με σαφή προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πώς θα γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα είπα ότι τις πρώτες 100 μέρες θα προσπαθήσουμε να βρούμε νέα οριζόντια νομοθεσία για τις δεοντολογικές και ανθρώπινες πτυχές της έχνης νομοσύνης. Παράδειγμα, θα μας ζητηθεί να δώσουμε περισσότερες ε, πληροφορίες. Ε, πρέπει να φροντίσουμε από την αρχή, από τον σχεδιασμό να γίνονται σεβαστά ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, από τον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας, μιας εφαρμογής ενός προϊόντος. Και θα πρέπει ακριβώς να κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις για τον αλγόριθμο και το σκεπτικό ε, από πίσω του, γιατί πρέπει όλες οι εθνικές αρχές και οι δικαστές να έχουν την ικανότητα να ελέγξουν. Οπότε με την Κομισιόν δεν σκοπεύουμε μόνο να νομοθετήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να οργανώσουν κάποιους ελέγχους για να λάβουν πληροφορίες. Βεβαίως θα υπάρξει νέα νομοθεσία, αλλά το έχω ήδη πει, θα εργαστούμε και κλαδικά, γιατί υπάρχουν ε, και άλλες ε, δυσκολίες στον ε, τομέα των μεταφορών και αλλού. Αυτό θα το συζητήσουμε λοιπόν με τους συναδέλφους, γιατί αν θέλουμε να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα, αν θέμε να μην υπάρξει διακριτική μεταχείριση, αυτό πρέπει να γίνει από τον σχεδιασμό ήδη. Γιατί δίνονται όλο και περισσότερες ε, προφορίες και πρέπει να δοθούν όχι μόνο στους καταναλωτές αλλά και στις αρχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια εμπειρία σας ε, στα ζητήματα εξωτερικών ε, και την δήλωσή σας ότι θέλετε έναν ισχυρό ρόλο στην εξωτερική διάσταση προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια θα είναι τα συγκεκριμένα βήματα που θα αναλάβετε για να προστατεύσετε το ευρωπαϊκό μοντέλο όπως ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πώς θα διασφαλίσετε πως οι διεθνείς διαπραγματεύσεις, ειδικά με τις ΗΠΑ, δεν θα υπονομεύσουν ε, την ε, προστασία αυτή του σχεδίου συμφωνίας και πώς θα φροντίσετε να αντέξει στα δικαστήρια. Και τέλος, θα επιβεβαιώσετε ότι με την Κομισιόν θα λάβετε μια ισχυρή θέση έτσι ώστε και στον τομέα της επιβολής του νόμου θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ε, και πάλι για την τελευταία σας ερώτηση, ε, ναι. Το, ε, απάντησα ναι. Η απάντηση είναι ναι για την δυνατότητα προώθησης ε, εκεί πέρα των προδιαγραφών μας. Ε, το είπα πολλές φορές. Αν θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, να πούμε ότι πολεμάμε την κλιματική αλλαγή, ότι προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εμελιώδεις αξίες. Αυτό πρέπει να γίνει όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε όλες τις συζητήσεις με τους διαφόρους εταίρους. Ε, μιλήσατε για τι είπα, Για να είμαι ειλικρινής, είναι και η Μπρίγκη Τζίπελ εδώ πέρα. Ε, εγώ είμαι ανοιχτό να καθίσω, να μιλήσουμε ε, για να δώσουμε στοιχεία, παραδείγματος χάνει, για να οργανώσουμε μια κοινή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να γίνει πριν ε, πάμε σε οποιαδήποτε συζήτηση με τη ΣΥΠΑ. Βεβαίω δεν σκοπεύω να ολοκληρώσω διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ πριν συμφωνήσουμε εντό τη Ένωση. Αλλά για να είμαι συγκεκριμένο, αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ε, θα έρθει η επιρροή από το εξωτερικό. Παραδείγματο χάρη νομοθεσία περί νέφου υπολογιστικού στις ε, ΗΠΑ. Έχει εξοδαφική εφαρμογή, οπότε πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε εμείς και να μην δεχτούμε επιρροή από έξω. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Μέλο από το ΕΛΚ. Κύριε Ρέιντερς, η κυρία Λάκοβέση θα είναι η νέα εισαγγελέα. Εσείς προβλέπετε άλλα μέτρα για ενίσχυση της θέσης αυτής κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Πιστεύετε ότι η Κομισιόν έχει κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκινήσει η λειτουργία της εισαγγελία το 2020 και ιδιαίτερα την ε, εφαρμογή της οδηγίας PIF που αποτελεί τη βάση για την εισαγγελία και επίσης ε, πρέπει να διασφαλιστεί επαρκές ανθρώπινο δυναμικό εγκαίρος. Και πώς μπορούμε Ε, να αποτρέψουμε επιδείνωση της ε, κατάστασης σε κάποια κράτη-μέλη, ε, ενθαρρύνοντας τα κράτη να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης, η πώληση ευρωπαϊκής ηθαγένειας ή διαβατηρίων, όπως γίνεται στη Μάλτα, Πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο, ιδιαίτερα όσον αφορά την νομοποίηση παράνομων εσόδων και τη φοροδιαφυγή. Και έληξε ο χρόνος σας, λέει η Πρόεδρος. So, thank you. First of all, Σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να επαναλάβω όσον αφορά την εισαγγελία ότι πρώτο έργο μας είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και έχω έρθει σε επαφή με τις παραμόδιες υπηρεσίες για να δω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Έχω λοιπόν ένα κατάλογο από πράγματα που πρέπει να κάνω μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες και έχω έρθει σε επαφή και με την κυρία Κοβέση ε, διότι είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε. Χρειαζόμαστε όμως καταρχάς ε, τη σώμα των επιτρόπων. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τα κράτη-μέλη και επίσης ε, πρέπει να φροντίσουμε για εφαρμογή της ε, οδηγίας PIF ε, διότι αλλιώς θα είναι δύσκολο να εργαστεί η νέα εισαγγελέα και επιπλέον θα είναι σημαντικό να διαθέσουμε σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους στη νέα εισαγγελία. Θα φροντίσω στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και από ό,τι φαίνεται έτσι είναι και η παρούσα ε, πρόταση. Ε, θα φροντίσω πάντως να υπάρχουν επαρκείς ε, πόροι για να γίνουν όλα αυτά. Μπορεί να είναι χρήσιμο να προχωρήσουμε και όσον αφορά την τρομοκρατία είπα ότι θα είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Δεύτερη ερώτηση, τα, ε, τα διαβατήρια. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει διευκόνηση και για κάποιες ε, τρίτες χώρες ε, όσον αφορά τις θεωρήσεις. Θα πρέπει να εμείνουμε στο πραγματικό δικό μας όραμα για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στο θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα Ε, Αποφασίστηκε να ε, δημιουργηθεί μια τέτοια ομάδα ε, που συγκεντρώνει σχετικές πληροφορίες. Είναι δύσκολο να έχουμε συγκεκριμένα νούμερα. Ε, με μια έρευνα λοιπόν θέλουμε να ασκήσουμε περισσότερη πίεση, να μάθουμε τον αριθμό των διαβατηρίων αυτών, ποιοι τα έχουν λάβει, διότι είπατε υπάρχουν κίνδυνοι διαφθορά, νομοποίηση παράνομων εσόδων και πολύ άλλοι κίνδυνοι. Είμαι διατεθειμένος λοιπόν να αγωνιστώ κατά αυτού, διότι πρέπει να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, συνδέεται με αξίες και ε, πραγματικά ελπίζω να μην δημιουργηθεί αγορά διαβατηρίων. Η ε, τήρηση του κράτους δικαίου είναι μια από τις ε, βασικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο περί δικαιοσύνης. Ε, είπατε ότι είσαστε προσιλωμένος ε, στην διεύρυνση όλων των εργαλείων δικαστικής συνεργασίας συμπεριλαμβανομένου του εντάλματος σύλληψης. Ε, όσον αφορά την παράνομη, τις παράνομες εκλογές στην Καταλωνία, η ε, πριν ε, δύο χρόνια ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κράτησε συγκεκριμένη θέση. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό και τέλος μετά από όσα ακούσαμε μέχρι τώρα από εσάς στηρίζετε τον τίτλο του χαρτοφυλακίου που επέλεξε η κυρία Φοντερ για το χαρτοφυλάκιο του Μαργαρίτη Σχοινά. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αυτό για μένα είναι το άρθρο 2 της συνθήκης. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Προστασία όλων των αξιών μας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό το έχω συζητήσει με την ε, εκλεγήσα πρόεδρο. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να εργαστούμε εργαζόμαστε, ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στο άρθρο 2 της συνθήκης και ε, θα επιμείνω για την άλλη σας ερώτηση στην θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να σεβόμαστε το, τη συνταγματική τάξη στα κράτη-μέλη. Αυτό το έχω πει και για το Βέλγιο, τη δική μου χώρα. Πρέπει να σεβόμαστε το, τη συνταγματική τάξη. Υπάρχουν κανόνε σε όλα τα κράτη-μέλη για αλλαγή της συνταγματικής τάξης, ε, αλλά θα εμείνω στη θέση αυτή. Και όσον αφορά το ε, ένταλμα σύλληψης, ε, αν χρειάζεται κάποια διαδικασία επιπαραβάση, αν χρειάζεται αναθεώρηση, θα το κάνουμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση είναι της κυρίας Κορνίλια Έρνστ από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η, η ερώτησή μου, κύριε Ράιντερς, είναι η εξή. Στην τελευταία ανακοίνωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του 2019, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται ως τομέας που θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Ε, είναι σημαντικό το θέμα της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και περιμένουμε από τον αρμόδιο επίτροπο να θέσει το θέμα αυτό ως προτεραιότητα στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβάσαμε όμως στον βελγικό τύπο ότι εσείς προσωπικά προτείνατε τροπολογία σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες ε, και φυλάκιση τριών ετών ε, ή ε, πρόστιμο 500.000 ευρώ. Κληθήκατε να τροποποιήσετε την πρότασή σας. Μπορείτε, παρακαλώ, να διευκρινίσετε τα περί αυτής της πρότασης. Ποια είναι η θέση σας και τι θα κάνετε εσείς ως Επίτροπος. Ευχαριστώ. Δύο ξεχωριστά στοιχεία υπάρχουν εδώ πέρα. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε διάφορους φορείς και διάφορες διαδικασίες στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Και είπα ότι θα προσαρμοστούν οι διατάξεις ανάλογα με τις προτάσεις αυτών των συμβουλευτικών ε, σωμάτων. Οι δημοσιογράφοι αντέδρασαν, ε, τους διαβεβαίωσα όμως ότι δεν σκοπεύουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητα ε, δημοσίευσης ε, κάποιων ε, πληροφοριών. Το πρόβλημα είναι για τους ανθρώπους που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. Δεν θέλουμε ε, να περιορίσουμε την ελευθερία του τύπου. Δεν ήταν αυτός ο στόχος ε, της νέας νομοθεσίας. Ως Επίτροπο σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να τεθεί σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία στα διάφορα κρατημέλη σχετικά με τις διαδικασίες ε, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Θα πρέπει να στήσουμε από τις εθνικές αρχές να επαληθεύουν τις πληροφορίες που δίδονται από τους ε, καταδότες δημοσίου συμφέροντος. Και από ψυχολογικής πλευρά είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Θέλω λοιπόν ως Επίτροπος να παρέμβω και να βεβαιωθώ να έχουμε πραγματική προστασία των πραγματικών μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Οι πολίτες ε, θα πρέπει να μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Υπάρχουν κάποια εχέγγυα. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι μιλάμε για πραγματικούς ε, whistleblowers, μάρτυρες ε, δημοσίου συμφέροντος. Θα εξετάσω την οδηγία και θα δούμε πως υπάρχουν νέα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε για να έχουμε καλύτερη προστασία τους. Κατάλαβα σωστά ότι θέλετε να αλλάξετε την πρότασή σας την πρόταση του καλοκαιριού. Θέλετε να αποσύρετε την πρόταση αυτή στο Βέλγιο. Κατάλαβα σωστά δηλαδή. Και η άλλη ερώτησή μου είναι... Ποια θέματα θα θέλατε, τι μέτρα θα θέλετε να λάβετε για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως δεν τα είπα καλά στα αγγλικά, στα πω γαλλικά, για να είναι πιο κατανοητό. Και στις ενώσεις ε, των Βέλγων ε, δημοσιογράφων και στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, που απευθύνθηκαν, τους δώσαν τεπάτσο, θα προσαρμοστεί το κείμενο με βάση αυτά που λένε και οι δημοσιογράφοι και το Συμβούλιο Επικρατείας και το κείμενο ε, ουσιαστικά θέλει να ορίσει τις περιπτώσεις όπου οι διαβασμένες πληροφορίες δεν μπορούν να διαδίδονται από τα άτομα που έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις πληροφορίες. Τελείως διαφορετική κατάσταση για τους δημοσιογράφους που φυσικά και δεν θέλουμε να πλήξουμε τα δικαιώματά τους. Ό,τι αφορά τώρα τους ίδιους τους καταγγέλλοντες, ε, φυσικά και πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία για τους προγραμματισμούς συμφέροντος παντού, αλλά ταυτόχρονα και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό με τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να εγκριθούν πληρωματικά μέτρα υποστήριξη συνδρομή. Αυτό θα μπορούσε να είναι δικαστική, νομική συνδρομή ή οικονομική συνδρομή. Επίση μπορεί να είναι και ψυχολογική υποστήριξη. Άρα σε όλα αυτά ε, με τα χαράς να δούμε πώς, μπορούμε, πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να πάνε πιο μακριά, αλλά και αν χρειάζεται να πάμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πιο μακριά. Μπόρζαν από τους ε, σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε από την ΙΜΚΟ ε, ένα σχόλιο. Είμαι λίγο απογοητευμένη γιατί το Mission Letter πολύ λίγα αναφέρει για την προστασία των καταναλωτών. Ελπίζω εσεί να εξασφαλίσετε ότι η προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη ευρωπαϊκών ε, πολιτικών και θα ληφθούν οριζοντίω ε, υπόψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει έναν πιο φιλοπεριβαλλοντικό σχεδιασμό για όλα τα προϊόντα και να είναι διαθέσιμα τα εξαρτήματα. Εμείς έχουμε ζητήσει τον ελάχιστο χρόνο ζωή, να είναι εγγυημένο και δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξη. Σε ό,τι διάφορα τη βιώσιμη κατανάλωση και την κυκλική οικονομία θα πρέπει για το ε, κύκλο των προϊόντων να είναι υπεύθυνοι κατασκευαστέ του. Ε, ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να έχουμε πιο βιώσιμοι τρόπου κατανάλωση. Συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για βιώσιμη κατανάλωση που να περιλαμβάνει την ευθύνη των παραγωγών, των κατασκευαστών. Ευχαριστώ. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβω και το είπα και στι αγωγέ μου παρατήρηση ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ε, τη ζήτηση για να ε, υπάρχει αυτή η ε, εξασφάλιση της κυκλικής οικονομίας. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης σίγουρα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Έχουμε τη Νέα Πράσινη Συμφωνία, τις πρώτες 100 ημέρες θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε ε, και με την πλευρά τη προσφοράς να εργαστούμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τώρα τους καταναλωτές θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν σε μια πιο ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία και είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη πληροφόρηση, πιο πολλά στοιχεία ενημέρωσης για τους καταναλωτές για να μπορούν να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές, επιλέγουν συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά δεν αρκεί αυτό όμως. Σε ό,τι διαφορά αυτή την πρόορη λήξη, ε, ημερομηνία λήξη, και επειδή έχω παραπλήσει πολλέ τέτοιε συζητήσει, πρέπει να προχωρήσουμε και όχι να ζητάμε θελοντικέ μόνο αντιδράσει. σω θα έπρεπε να σκεφτούμε αν μπορούμε νομοθετικά να αντιδράσουμε για να πάψει να ισχύει αυτή η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξη. Να συζητήσουμε επίση τη βιωσιμότητα, ε, τη διάρκεια ζωή των προϊόντων και να μπορεί κανείς να ε, ζητά από τι εταιρείε να δίνουν πληροφορίες για τη βιωσιμότητα, για τη δυνατότητα επισκευή, για τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων ανταλλακτικών. Τέλος πάντων, ε, καλή πληροφόρηση προς τους ε, καταναλωτές. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την ευθύνη, επειδή μιλήσατε και για την ευθύνη, ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να υπάρχει ενημέρωση για να επηρεάσει ε, αυτό την ευθύνη των καταναλωτών. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρη, δηλαδή να αναφέρεται ξεκάθαρη διάρκεια ζωής του προϊόντος και δυνατότητα επισκευής, να είναι εγγυημένη και το greenwashing είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγουμε και πρέπει να υπάρχει πραγματική πληροφορία, όχι παραπληροφόρηση ή ψευδείς ειδήσει ε, που κάποιες φορές δίνονται στους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Άκουσα ε, τι είπατε στην εισαγωγική σας ομιλία κυρία Μπόρζαν. Απλά θα ήθελα και γραπτός να τα δω. Και κάτι τελευταίο στις ειδήσει πρόσφατα αναφέρεται ότι έχουμε ε, πολύ μεγάλες αυξήσεις στις εισαγωγές ηλεκτρικών συσκευών, για παράδειγμα, από τρίτες χώρες ε, που μπαίνουν ε, στην ευρωπαϊκή αγορά της ΥΟΣ και τα πρώτα αυτά δεν είναι πάντοτε ασφαλή προς χρήση από τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών από μη συμμορφούμενα αγαθά στην Ευρωπαϊκή Αγορά και ακόμη περισσότερο. Πώς θα βοηθήσετε ώστε η ενίσχυση της τουρκικής αγοράς να μην μειώσει τα επίπεδα προστασία ε, των καταναλωτών. Και δεν έκανα καν ένα λεπτό, ε. Συγχαρητήρια, λέει ο κύριο Ρέντες. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Είπα ένα για τις διαδικτυακές πωλήσει στο e-commerce. Εκεί μπορούμε να συνεργαστούμε με τις πλατφόρμες και να ζητάμε από τις πλατφόρμες να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο για τα παράνομα προϊόντα, όπως είπαμε, αλλά και για προϊόντα που έχουν ρίσκο, Δεν έχουν ρίσκο, ε, κίνδυνο αφού γίνει η ανάλυση κινδύνων, αν υπάρχει κίνδυνο, θα πρέπει να ε, αφαιρούνται από την πλατφόρμα. Και με την Κίνα, για αυτό σαν ένα παράδειγμα. Στις συνομιλίες μας θα τους πούμε ότι θέλουμε να εξάγουν ασφαλή προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν αφορά ε, το ψηφιακό κόσμο, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Πρέπει να πούμε ότι μια αλλαγή, μια αναθεώρηση ίσως του δικτύου ασφαλεία, τη γενική προστασία που έχουμε για την ασφάλεια των ε, προϊόντων, ίσως χρειάζεται να αλλάξει σχετική οδηγία, αλλά τέλο πάντων, από όλε αυτές τις πιθανές δράσεις, σίγουρα αυτό που πρέπει ε, προτεραιότητα να έχει είναι η έλεγχη των πρώτων που έρχονται στην Αστική αγορά. Να ερευνάτε ο κίνδυνο για την ασφάλεια και αν υπάρχει κίνδυνο πρέπει να αντιδρούμε. σω αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο, μάλλον ίσω ο καλύτερο τρόπο γι' αυτό είναι να αναθεωρήσουμε το ΔΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων. Και όχι μόνο με ένα γενικό δίκτυο ασφαλεία, αλλά ίσω ανακλάδο, ανατομέα, να υπάρχουν διαφορετικοί ε, κανόνε εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ευχαριστώ. David Corman από του Πρασίνου Merci, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε υποψήφια επίτροπε. Άκουσα την απάντηση που δώσατε στη συνάντηση και την ευχαριστώ που έθεσε την ερώτηση για την υπεύθυνη ε, βιώσιμη κατανάλωση. Βέβαια, η απάντηση δεν μας ικανοποιεί. Ε, τέλος. Λέτε ότι πρέπει να δείξει υπευθυνότητα ο καταναλωτής, αλλά η υπευθυνότητα και ευθύνη των βιομηχάνων, γιατί εκεί είναι το θέμα. Αν είμαστε νομοθέτες, ε, δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε τις καλές συμβουλές στους καταναλωτές, αλλά για να νομοθετούμε. Και κάθε σοβαρή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της προγραμματισμένης μερομηνίας λήξης και της βίωσης κατανόησης, θα πρέπει να ορίζει νέα πρότυπα, θα πρέπει να ε, κάνει τους παραγωγούς να εγγυώνται την ποιότητα, την ε, διάρκεια ζωής, τη βιωσιμότητα προϊόντων. Και η νόμη εγγύηση επίσης που είναι δύο χρόνια. Θα το ξαναδείτε, θα δείτε την οδηγία σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών για να αυξήσετε την εγγύηση σας στα 5 ή 10 χρόνια, ώστε να είναι εγγυημένη η ευρωστία προϊόντων και τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα να είναι διαθέσιμα. Και τι θα γίνει με την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξη, αν δεν γίνονται σεβαστά ε, τα σχετικά, θα επιβάλλετε κυρώσει ε, και τι θα κάνετε με τι επιχειρήσει για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Ε, Σα ευχαριστώ κύριε Κόρμα. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη κατανάλωση και τη διάρκεια ζωής. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να δίνουν σωστές πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη αυτά τα οποία είπατε, τη διάρκεια ζωής, ε, τη δυνατότητα επισκευής, ε, επιδιόρθωση και τη διάθεση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Και επισκευή ίσως και από τρίτους, όχι απλά μόνο από την επιχείρηση. Άρα, για όλα αυτά, βεβαίως και μάλλον θα χρειαστεί να νομοθετήσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι υπάρχει συγκεκριμένα, ποιες είναι οι διατάξεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά αν θέλουμε να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει φυσικά να υποχρεώσουμε τους παραγωγούς να δίνουν αυτές τις πληροφορίες και να εγγυώνται. Να εγγυώνται. Είπατε για την εγγύηση, αν θα πρέπει να ε, επιμηκυνθεί. Θα το εξετάσουμε, είμαι ανοιχτό. Θα εξετάσουμε όλες τις υποθέσεις για να δούμε κατά πόσον ε, υπάρχει δήλωση τη διάρκεια ζωή, θα πρέπει να είναι και εγγυημένη. Είναι λογικό αυτό. Θα είναι 5 ή 10 χρόνια εγγύηση. Ε, είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Σε εδώ, ό,τι διάφορα την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξη. Αν είναι προγραμματισμένη, αυτό σίγουρα θα πρέπει να θεωρηθεί παράβαση και να μπορούν να επιβληθούν κυρώσει σε επιχειρήσει που το κάνουν. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνει αυτή η λογική ε, εκούσια ε, της προγραμματισμένης μερομήνας λήξης και να μην τιμωρούμε αυτούς που το κάνουν. Και φυσικά και πρέπει να κινητοποιήσουμε τους καταναλωτές για να ενημερωθούν, αλλά θα πρέπει, δεν αρκεί αυτό, θα πρέπει να υποχρεώσουμε τους ε, κατασκευαστές, τους παραγωγούς να βάζουν στοιχεία για τη διάρκεια ζωής, να τότε επισκευής και από τρίτους, ε, ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αν χρειαστεί να τιμωρούμε την προγραμματισμένη ημερομηνία Του Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι ε, πρόωρα ε, πάβει να λειτουργεί ένα προϊόν που θα μπορούσε να λειτουργήσει για πιο πολύ χρόνο. Φυσικά και θα πρέπει να νομοθετήσουμε από αυτό και να δούμε πώ πρέπει να ε, ενισχύσουμε την ευθύνη και των παραγωγών. Ο κύριο Κορμά, ευχαριστώ. Επανέρχομαι στο έρθμα τη κυρία Έρνστ για του μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο. Δεν κατάλαβα πολύ καλά όλη σας την απάντηση. Σαν ε, ε, Δόκτωρ Ρέιντερς και Μίστερ ε, Didier μας τάπατε. Τι θέλετε να κάνετε για να ενισχύσετε τα δικαιώματα και την προστασία των καταγγελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που συχνά ξέρετε ότι είναι το πρώτο όπλο κατά τον λόμπι που καταγγέλουν, έχουν το στένος να καταγγείλουν αξιόπινες πράξεις. Ανησυχώ γιατί εσείς αναλάβετε τη δικαιοσύνη και την πραγματική προστασία των ηρώων αυτών της σύγχρονης εποχής, που είναι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Απάντηση. Παναλαμβάνω. Έχουν προσαρμοστεί στο Βέλγιο τα κείμενα με βάση τα αιτήματα των ενώσεων των δημοσιογράφων και του ε, Συμβουλίου Επικρατεία. Ε, κλασικά έτσι γίνεται στη χώρα μας. Τα κείμενα δηλαδή θα είναι σύμμορφα προς όσα έχουν πει οι ίδιε οι ενώσει των δημοσιογράφων στου οποίου συμβουλευτήκαμε. Δεύτερον, για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα διαβεβαίω, ανεξαρτήτως των δικών προσωπικών εμπειριών, εγώ θέλω να είναι εγγυημένη η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμμετοχή. Τι θα πει αυτό ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει πραγματική εφαρμογή τη οδηγία. Η οδηγία υπάρχει. Θα πρέπει να εφαρμόζεται. Σήμερα δεν συμβαίνει παντού αυτό. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε λοιπόν και μπορούμε να φτάσουμε και σε διαδικασίε επί παραβάση. Τώρα, αν κάποια κράτη θέλουν να πάνε πιο πέρα, πώ μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του, ε, μπορούμε να του βοηθήσουμε αυτά τα κράτη και να δούμε ίσω και με, την, ε, με, την, ε, με το θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν τέτοια δείγματα. Φυσικά, βέβαια, θα πρέπει να είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχουν και πραγματικού καταγγέλλοντε στην οδηγία. Υπάρχουν ρήτρε διασφάλιση, αυτό μου φαίνεται προφανέ. Γιατί αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να υπάρχουν τέσσερι ρήτρε. Άρα, κανένα πρόβλημα και καμία αμφιβολία. Ναι, θα προσχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα έχουμε καθυστερήσει. Παρακαλώ, δύο τελευταίε ερωτήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομε. Έχετε τον ε, λόγο, κύριε Σένμακερ, από το Ρήνιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και κύριε Ράιντερ που ήρθατε και απαντήσατε στις ερωτήσεις. Ήδη ανέπτυξα κάποια στοιχεία για τις ε, μικρομεσαίες και τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις και θα ήθελα να σας πω πως ε, θα έχουμε μια νέα εξέλιξη στην οικονομία με όλο και περισσότερο ψηφιακή προσέγγιση που μας δίνει μια πάρα πολύ ευκαιρία για να υπερασπιστούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις startup. Η οδηγίες για το θέμα αυτό, την ψηφιοποίηση δηλαδή του εμπορικού δικαίου μας δίνει κάποιες δυνατότητες. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε παραδείγματος χάρη το ψηφιακό ως την πρώτη επιλογή, τη φυσική επιλογή, με λιγότερο χαρτί, με λιγότερη γραφειοκρατία, να έχουμε ως πρώτο σημείο αναφοράς την ψηφιακή προσέγγιση. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σε κάθε ε, νέο κανόνα που θα τίθεται ενισχύ, όπως παραδείγματο χάρη είναι η νομοθεσία για την τεχνητή νομοθεσία. Ε, συγγνώμη. Ε, όχι, α το πω αγγλικά. απλά να πω ότι θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να δούμε τις διάφορες ιδιαιτερότητες στους ε, κανόνες για τις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Μίλησα για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην φροντίσουμε λοιπόν όπως ε, και στην προστασία δεδομένων έχουμε συγκεκριμένους κανόνες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νέοφυής ε, είπατε μια ειδική άδεια για αυτέ τι επιχείρησει είναι μια καλή ιδέα. Πρέπει να το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για να έχουν κάποιο είδου διαβατήριο να δουλέψουν σε άλλε χώρε, Ε, παίρνοντας ένα τέτοιο διαβατήριο από μια χώρα βεβαίω είμαι υπέρ. Ε, γιατί το έχουμε και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών. Γιατί όχι λοιπόν, αν θέλει κάποιο να επενδύσει στην καινοτομία. Θα το κάνουμε λοιπόν αυτό και να σκεφτούμε του ίδιου κανόνε για τι μικρομεσαίε ε, επιχείρησει. Αυτά λοιπόν για να ολοκληρωθεί η συζήτηση σε δύο γλώσσε. Ευχαριστώ για την απάντηση και σα ευχαριστώ για αυτά τα θετικά τα οποία είπατε για την άδεια. Για την ψηφιοποίηση υπάρχει κάτι άλλο που είναι εμπόδιο στις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Είναι τα πολλά δεδομένα που παραμένουν στι ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι αναγκαίο για πολλέ ε, επιχειρήσει. Ακριβώ να έχουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να καινοτομήσουν. Τι άποψη έχετε λοιπόν για τα δεδομένα business to business ε, μεταξύ των επιχειρήσεων. Ε, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την ιδιοκτησία αυτών των δεδομένων για να προωθηθεί η καινοτομία και επίσης σημαντικό τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα είναι ε, ίσως κάτι το οποίο θα κάνει η Κομισιόν τις πρώτες εβδομάδες να υπάρξει αυτή η ισορροπία στην προστασία της ιδιωτικότητας κάποιων ε, δεδομένων ε, στην δυνατότητα να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και από την άλλη να προωθήσουμε την ε, καινοτομία και να υπάρχει να υπάρχουν ακριβώς τα απαραίτητα δεδομένα για να προωθεί αυτή η καινοτομία. Όπως είπα θα δούμε πώς θα καταστεί δυνατόν συγκεκριμένα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι, όπως είπα, αν ζητάμε όλο και περισσότερες ε, πληροφορίε από του καταναλωτές ε, στις σχέσεις ε, μεταξύ επιχειρήσεων, θα πρέπει να δοθούν και περισσότερες πληροφορίες για το πώς διαχειρίζονται τη χρήση τεχνητή νοημοσύνης εντό τη επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί η, η, η ισορροπία αυτή π.χ. μεταξύ της πνευματικής ιδιοκτησίας μιας εταιρείας και της πρόσβασης άλλων εταιρείων. Θα πρέπει λοιπόν τις πρώτες ε, εβδομάδες να δούμε την διοντολογική προσέγγιση και την ανθρώπινη προσέγγιση της ε, τεχνητής νομοσύνης αλλά και την προσέγγιση αυτή της ιδιωτικότητας με καινοτομία την ιδιωτικότητα με την ανάγκη να μοιραστούν αυτές οι πληροφορίε για να μπορέσει να προωθηθεί η καινοτομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Βάουτσμαν από το ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Ράιντερς, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα κλείσω τη σειρά αυτή των ερωτήσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις σαφείς ε, απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ε, ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει και σε μια καλή συνεργασία. Συμφωνώ ότι ε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιστημονική φαντασία. Ήδη σήμερα ε, είναι πραγματικότητα στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι απαραίτητες οι διατομεακές λύσεις ε, και στις γραπτές σας απαντήσεις. Αναφερθήκατε στη διοντολογική πλευρά, αναφερθήκατε και στην προστασία των δεδομένων. Έχω την εξής ερώτηση. Έχετε σκοπό μέσα στις πρώτες 100 μέρες να υποβάλλετε πρόταση ε, για την ευθύνη των προϊόντων ε, τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή όχι τροποποίηση παλιάς, ε, παλιάς νομοθεσίας, αλλά νέα νομοθεσία για το θέμα αυτό. Ίσως θα πρέπει να το διευκρινίσω αυτό. Όχι. Δεν είπα ότι θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο σε, δυνατό σε, στις πρώτες 100 μέρες. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες, όπως είπε και η εκλεγήσα πρόεδρος ε, κυρία Φοντερ Λάιεν, θα εκπονήσουμε μια προσέγγιση για τον ψηφιακό κόσμο, ε, έχοντας κατά νου ιδιαίτερα τις ε, δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου με το χαρτοφυλάκιο αυτό, θα ασχοληθούμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει οριζόντια προστασία και θα πρέπει να σκεφτούμε τις δεντολογικές και ανθρώπινες πτυχές. Ε, με τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες ε, θα πρέπει να εξετάσουμε την ευθύνη των προϊόντων και είπα στον ε, κύριο Πέτερς για τα... μίλησα στον κύριο Πέτερς για τα αυτοκίνητα που θα έχουμε χωρίς οδηγούς ε, ποιος θα είναι υπεύθυνο σε περίπτωση ατυχήματος ο ιδιοκτήτης, δεν υπάρχει οδηγός, η επιχείρηση, η εταιρεία ε, που δημιούργησε τον αλγόριθμο θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες ε, γνωρίζω ακριβώς τι θα κάνω, διότι είναι πολύ αναλυτική η επιστολή ανάθεσης καθηκόντων μου. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα όσον αφορά την ευθύνη. Είπα ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με την ευθύνη για τα προϊόντα, ε, διότι μας ενδιαφέρει η ασφάλεια. Ε, έχουμε μετά τις διοντολογικές ηθικές πτυχές, ε, αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι μέσα στις 100 πρώτες μέρες θα έχουμε νέα πρόταση για την ευθύνη των προϊόντων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τότε να ρωτήσω το εξής. Εγώ είμαι τακτικό μέλος και της Επιτροπής ε, για τη Δικαιοσύνη και για την Εσωτερική Αγορά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η οριζόντια προσέγγιση στην νομοθεσία. Δεν είναι όμως ε, πάντα πολύ ε, εύκολο να λαμβάνουμε υπόψη όλους τους τομείς. Ε, θα είναι λέξη generalis, γενικός νόμος, η οριζόντια νομοθεσία και θα προβλέπετε λέξη specialis, ειδική νομοθεσία για τους διάφορους τομείς. Και τι, τι σκοπεύετε να κάνετε πρώτα. Ακούστε η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν μας εμπιστευτείτε, θα είναι ότι ευθύς εξ αρχής να υπάρχει οριζόντια νομοθεσία για τις ανθρώπινες και ηθικές πτυχές. Αυτή θα είναι η προσέγγιση και το λέω όχι για τους χρήστες μόνο, αλλά και για τις αρχές ελέγχου και για τις, ε, τα δικαστήρια που θα πρέπει να αποφανθούν. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες ε, και στο τι γίνεται γενικώ στον τομέα της τεχνητής δικαιοσύνης και όπως είπα, στους τομείς όπως είναι μεταφορές, η υγεία, η ε, χρηματοπιστωτικός κλάδος, εκεί θα πρέπει να δούμε μήπως χρειάζεται πιο ειδική συγκεκριμένη λεπτομερής προσέγγιση. Και αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τους αρμοδίους ε, επιτρόπους. Η ευθύνη για την ευθύνη ίσως να είναι η ίδια προσέγγιση. Δηλαδή να έχουμε ένα προσαρμοσμένο σύστημα, αλλά μετά να εμβαθύνουμε τομέα ενδεχομένως. Άρα στα δύο επίπεδα που λέτε θα εργαστούμε πράγματι. Σα Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές και για τις ερωτήσεις και για τον Επίτροπο για τις ε, απαντήσεις του και τώρα θα σας δώσω το λόγο για μια καταληκτική παρέμβαση, πέντε λεπτά. Ο κύριο Ρενιντές, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ, πρώτα απ' όλα θέλω να σα ευχαριστήσω για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων που έρχεται ω συνέχεια των διαφόρων ανταλλαγών απόψεων. Προσπάθησα να έχω με μέλη τη Επιτροπή σα τέσσερις εβδομάδες. Ξέρω ότι κάποιες φορές είναι ζωντανέ, έντονε οι ανταλλαγές αυτές απόψεων. Το ίδιο ε, και στην εθνική, σε εθνικές ε, ε, Συνελευσει ε, είναι έντονε αυτές οι συζητήσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ε, ότι προσπάθησα να σα δώσω κάποιες βασικές γραμμές, σεβασμό κράτο δικαίου, δικαιοσύνη, προστασία καταναλωτών. Αυτά είναι τα τρία σκέλη του χαρτοφυλακίου μου. Σήμερα στην παρέμβασή μου προσπάθησα να σα παρουσιάσω τις προτεραιότητε που έλαβα και στο Mission Letter, την επιστολή ανάληψη καθηκόντων μου, αλλά δεσμεύομαι να ε, κάνω να προοδεύσω τα πράγματα στο θέμα ε, του κράτους δικαίου. Το σημαντικό μας ήταν να σας ακούσω ταυτόχρονα και να νιώσω και τι σας ανησυχεί γιατί θα εργαστούμε από κοινού. Ξέρω πώς λειτουργεί το Συμβούλιο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να έχει ε, την υποστήριξη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να καταθέσουμε νέες πρωτοβουλίες. Εγώ αυτή τη φιλοδοξία έχω τουλάχιστον και αυτό ζήτησε και η κυρία Φοντρελάνη για το δικαίωμα πρωτοβουλία. Συνεχίζω λοιπόν να προωθώ τις προτεραιότητες αυτές, να προασπίσω εφαρμόζουν το κράτο δικαίου στα κρατημέλη και στι χώρε γειτονία. Θέλω να υπάρξουν επίση νέοι μηχανισμοί για το κράτο δικαίου. Επίση, τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να τύχουν πλήρου προστασία στην ψηφιακή εποχή, όπω είπαμε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί. Θέλουμε επίση να έχουμε μια δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων, να λάβουμε πρωτοβουλίε στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνη, να ενθαρρύνουν του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει να κάνουν επιλογέ βιώσιμε, να ενισχύσουμε τι δυνατότητε ε, συλλογική Ένωση προστασία και να εγκριθεί γρήγορα και η οδηγία για τι ε, δράσεις αντιπροσώπευσης για να προστατεύσουμε τη ελευθερία κυκλοφορία επίση των πολιτών ε, στο πλαίσιο και του Brexit που είναι ακόμη πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Κάτι ε, άλλο το οποίο συζητήσαμε ε, και νομίζω, μάλλον πολλά άλλα θέματα τα οποία αναφέρατε, θα τα λάβω υπόψη μου και ελπίζω να μπορέσουμε να τα ανταμετωπίσουμε όπως και αυτά που θα ανακύψουν στην επόμενη πενταετία. Ε, λίγες μόνο εβδομάδες ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ μας και συνεχίστηκε και σήμερα και είμαι διατεθειμένος να τον συνεχίσω αυτό το διάλογο. Θα σας συναντώ σε τακτά διαστήματα όποτε εσείς κρίνετε ότι είναι απαραίτητο και νομίζω ότι ε, χρήσιμο θα ήταν να έρχομαι στον τον πιο συχνά συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι θα υπάρξουν εμπόδια, το ξέρετε κι εσείς, δεν είναι εύκολο οι συνομοθέτες να συμφωνήσουν, όμως ε, να είστε βέβαιοι ότι εγώ είμαι αποφασισμένος και θα προσπαθήσω να το πετύχω αυτό. Και ολοκληρώνοντα να πω ότι ευτυχώ δεν μιλήσαμε για την ε, τεχνητή νοημοσύνη υπό την έννοια ότι υπάρχουν μαύρα ε, σημεία ε, υπήρξε ένα μαύρο σημείο σήμερα που ήταν το blackout που πάθαμε, αλλά άλλα blackout δεν υπήρξαν και θέλω να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις ε, που μας βοήθησαν ε, και μπορέσαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Thank you very much indeed, Commissioner. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για τις ε, πάρα πολύ χρήσιμες ε, και ε, απαντήσεις σας και τη σύντομη σας δευτερολογία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτέ και για τις ερωτήσεις αλλά και για την συνεργασία και την υπομονή που δείξατε επειδή χρειάστηκε να αλλάξουμε αίθουσα. Ευχαριστώ και δίνω στον πρόεδρο της Επιτροπής Λίμπε το λόγο για να κλείσουμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ελευθεριών ε, Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις ε, και ειδικά τον κύριο Ρεντέρς για την ενέργεια που επέδειξε και την υπομονή σας. Ξεπεράσαμε το αναπάντεχο αυτό περιστατικό, το σλιβερό αυτό blackout αλλά ε, κρατήσατε τεταμένη την προσοχή της αίθουσας. Ε, προσέλευση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πριν από τέσσερις ώρες. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές. Ε, πραγματικά όλοι κρεμόταν από τα χείλη σας. Γιατί βεβαίως είναι πάρα πολλά τα θέματα του σας, δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, προστασία των καταναλωτών ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στην επόμενη εντολή της ε, Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ε, και για τον χρόνο σας, για την υπομονή σας και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεργασία σας, ε, για την κατανόησή σας στην σημερινή συνεδρίαση. Just an The coordinators... Οι συντονιστές θα συνεδριάσουν σήμερα μία με δύο η ώρα το μεσημέρι η μικτή επιτροπή αξιολόγησης από τις επιτροπές Γιούρι, Λίμπε και Ίμκο επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.